Αρχίζουμε. Έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Κυρία Μπιλμπάου, θέλετε κάτι να πείτε, βλέπω. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Πρόεδρε, θα ήθελα να σας πω ότι έρχομαι από άλλη ψηφοφορία από την Επιτροπή Ελίας. Άφησα την ε, κάρτα μου εκεί. Θα σηκώνω το χέρι για να δείτε πώς ψηφίζω, έτσι. Την ξέχασα εκεί την κάρτα μου, την ηλεκτρονική. Και εσείς, κύριε Ρικέ, το ίδιο πρόβλημα. Το κατάλαβα. Αρκεί να μου χαμογελάσετε. Σηκώνετε το χέρι ευκρινώς για να μετρηθεί η ψήφο σας. Αρχίζουμε κάνοντας μία πρόβα, ένα τεστ, να δούμε αν έχουμε παρτία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Πολύ ωραία. Αρχίζουμε τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών. Αρχίζει η ψηφοφορία. Α, βρήκε η κυρία Μπιλμπάου την κάρτα της, κύριε Ρικέ. Λίγη ψηφοφορία. Ομόφωνα εγκρίθηκε η έκθεση αυτή. Ψηφίσατε υπέρ. Άρα είμαστε 43 υπέρ. Εντάξει, πολύ ωραία. Περνούμε αμέσως στην ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Μάια Μάρκοβιτς Κοστελάκ, εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στην Θάλασσα. Είναι εδώ η κυρία Κόστελακ. Σας καλωσορίζουμε κυρία Κόστελακ. Merci beaucoup. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Με ευχαρίστηση υποδεχόμαστε στην Επιτροπή μας την κυρία Μάρκοβιτς Κοστελάκ, εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Μετά από τις εκλογές του 2019 είχα αποφασίσει ότι θα καλέσω τους διευθυντών στους εκτελεστικού διευθύντε των τριών ευρωπαϊκών οργανισμών που μα εκπροσωπούμε και θα ήθελα να καλωσορίσω την ε, εκτελεστική διευθύντρια που άρχισε την θητεία της την 1η Ιανουαρίου φέτος, την επισκεφθήκαμε το Φεβρουάριο, πάντα είχαμε με την ε, πάρα πολύ καλή συνεργασία και θα θέλαμε να μας μιλήσετε για τις δραστηριότητες και τα επιτεύγματα του οργανισμού σας και τι προβλέπετε να κάνετε στο μέλλον, διότι όπως ξέρετε οι θαλάσσιες μεταφορές είναι και θέμα που μας υποσχολεί ιδιαίτερος. Για έξι λεπτά, κυρία Μάρκοβιτς, έχετε το λόγο και μετά συμμετέχετε στην συζήτηση. Θα μιλήσετε αγγλικά. Πολύ ωραία. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, ε, πραγματικά είναι χαρά για μένα το ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ για δεύτερη φορά ε, το 2019. Είναι η πρώτη φορά που μου δίνεται ευκαιρία να σας παρουσιάσω την ΕΜΣΑ στην Επιτροπή και επίσης ε, να μπορέσω να σας παρουσιάσω τη στρατηγική ε, πέντε ετών που έχουν χαράξει. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι θαλάσσιες μεταφορές είναι καθοριστική σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ε, σε ολόκληρο τον κόσμο πάνω από το 80% του εμπορίου αγαθών ε, γίνεται μέσα από θαλάσσιες μεταφορές και το ίδιο ισχύει και σε διεθνές επίπεδο. Περίπου το 33% του ενδοενωσιακού εμπορίου γίνεται μέσα από ευρωπαϊκά λιμάνια. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικός παίκτη ε, σε διεθνές επίπεδο. Έχει περίπου το 40% του παγκόσμιου θαλάσσιου τονάζου. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει αυξηθεί το εμπόριο στις θαλάσσιες μεταφορές και αυτό συμβαδίζει και με το ότι αυξάνεται και ο όγκος και η πολυπλοκότητα της ναυτιλίας. Παρότι λοιπόν υπάρχουν αλλαγές, παρόλα αυτά θεωρώ ότι μπορούμε να πούμε με άνεση ότι αυτή τη στιγμή η ναυτιλία βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Έχουμε τις ε, τεχνολογικές εξελίξεις που αλλάζουν τις ε, καθημερινές μας δραστηριότητες και εδώ θα έλεγα ότι επικρατεί όλο και περισσότερος αυτονομισμός ε, και έχουμε απόλυτα αυτόνομα σκάφη. Σε συνδυασμό με τα νέα μεγάλα σκάφη όπως γνωρίζετε όλα αυτά θα αλλάξουν τη ναυτιλία και υπάρχει δυνατότητα σε μεγάλο βαθμό να περιοριστεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των θαλάσσιων μεταφορών. Εξάλλου υπάρχει ευκαιρία για οικονομική ε, ανάπτυξη με βάση εφής λύσεις και την χρήση της ε, τεχνολογίας. Όμως, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όλα αυτά δεν προκύπτουν ε, χωρίς προβλήματα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην ασφάλεια ε, και στην σταθερότητα σε επίπεδο κοινωνικό. Εμείς είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε ε, στις ε, προκλήσεις, ε, όλα αυτά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, μπορούμε να κάνουμε τη βέλτιστη χρήση των πόρων μας. Σε θεσμικό επίπεδο έχουμε τώρα ένα νέο κοινοβούλιο, μια νέα επιτροπή, νέες προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΜΖΑ συμβάλλει χειροπιαστά σε όλα αυτά. Έχουμε ένα νέο PDP το οποίο θα τεθεί θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2021 και αυτή τη φάση, σε αυτή τη φάση είμαστε σε διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, σας είμαι ευγνώμων που δέχεστε το αίτημά μας να έχουμε ένα σταθερό προϋπολογισμό και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσετε να μας στηρίζετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν λοιπόν ε, σας ε, παρουσιάσω τη νέα μας στρατηγική, επιτρέψτε μου σύντομα να σας παρουσιάσω τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Ε, συστήθηκε το 2 στα πλαίσια του πακέτου ΕΡΙΚΑ 2 ως απάντηση στις μεγάλες καταστροφές των τάνκερ Έρικα και Πρεστίζ που ρήπαναν εκατοντάδες χιλιόμετρων των ακτών μας. Ο κανονισμός που μας ε, Διέπει, έχει αλλάξει αρκετές φορές, τελευταία φορά το 2016, έτσι ώστε η ευρωπαϊκή συνεργασία ε, για θέματα ε, ακτογραμμής να ενταχθεί και αυτή στις αρμοδιότητές μας. Με βάση λοιπόν τον ε, κανονισμό περί χρηματοδότησής μας, εμείς είμαστε αποκεντρωμένος οργανισμός, ε, συστήθηκε ο οργανισμός μας ε, για να έχουμε ένα αποτελεσματικό επίπεδο θαλάσσιας ασφάλειας, πρόληψη στη ρήπανση που προκαλείται από σκάφη και επίσης στόχος μας είναι να ε, αντιμετωπίσουμε και την ε, θαλάσσια ρήπανση που προκύπτει από όλες τις εγκαταστάσεις αερίου, που χρησιμοποιούν αέριο. Με βάση τον κανονισμό χρηματοδότησης, η ΕΜΣΑ πρέπει να τα επιτύχει όλα αυτά, προσφέροντας τα κράτη-μέλη και στην Επιτροπή τεχνική και επιστημονική υποστήριξη και υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, έτσι ώστε να εφαρμόζεται η ενωσιακή νομοθεσία, να ε, είναι εύκολο να ελέγχεται ελέγχονται οι πράξεις μας, όλα αυτά τα οποία αποφασίζουμε. Η ΕΜΣΑ έχει επίσης και μία σειρά επιχειρησιακών καθηκόντων. Έχουμε μία εργαλειοθήκη για να βοηθούμε τα κρατημέλη να αντιμετωπίζουν τη ρήπανση και επίσης ε, και ε, για να υπάρχει καλύτερος έλεγχος. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε και drone. Οι πόροι μας αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε περίπου 83 εκατομμύρια ευρώ. Ε, το Διοικητικό μας Συμβούλιο αποτελείται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την Νορβηγία, την Ισλανδία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε 270 ιδιαίτερα καταρτισμένους υπαλλήλους. Από το 6 βρισκόμαστε στη Λισαβόνα, εκεί είναι η έδρα μας. Η πλειοψηφία του προσωπικού μας ε, έχει γνώσεις ε, σε θαλάσσια θέματα και πρέπει να γνωρίζετε όλοι ότι ε, έχουμε 36% γυναικών, κυρίως βέβαια άνδρες, και θα ήθελα το ποσοστό των γυναικών να αυξηθεί περισσότερο, να φτάσουμε μέχρι το τέλος της θητείας μου σε 50-50% εκπροσώπηση. Όλα αυτά να συμβαδίζουν με τις ε, με, την, με, την, ε, με τον καταμερισμό στο διοικητικό συμβούλιο που είναι εννέα, ε, με συγχωρείτε, τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες. Έχουμε την επιτροπή, την της επιτροπή μεταφορών που είναι γυναίκα. Εγώ είμαι γυναίκα. Έχουμε την ε, γυναίκα νέα πρόεδρο της επιτροπής, άρα πράγματι έχει σημειωθεί ε, πρόοδο σε θέματα μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι ένα ε, χειροπιαστό παράδειγμα για το πώς στηρίζουμε τις γυναίκες ε, να εξελιχθούν στον τομέα των μεταφορών. Να δούμε τι ακριβώς κάνουμε στην ΕΜΣΑ. Εμείς, όπως σας είπα, στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, θεσπίζει νέα ε, νομοθεσία, να υπάρχει εναρμόνιση στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής με την διεθνή νομοθεσία. Πρόκειται να κάνουμε 22 επισκέψεις στα κράτη-μέλη, 16 επισκέψεις αναγνωρισμένων οργανισμών και ελέγξαμε 5 αποκαλούμενες τρίτες χώρες για το κατά πόσον πράγματι είναι ε, νομότυπα τα πιστοποιητικά τους. Φέτος ε, θα εξετάσουμε το θέμα των ε, πυρκαγιών Επίσης θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα σκάφη κάνουν τις μανούβρες και τα αυτόνομα σκάφη. Προσφέρουμε τεχνογνωσία στο προσωπικό μας, ε, εναρμονισμένη τεχνογνωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρυσι είχαμε πάνω από χίλιους υπαλλήλους που παρακολούθησαν την εκπαίδευση, χρησιμοποίησαμε την τελευταία τεχνολογία και ε, εργαλεία εκμάθησης εξ Χρησιμοποίησαμε και την εικονική πραγματικότητα. Αναπτύσσουμε εργαλεία για να στηρίζουμε τις επιθεωρήσεις των σκαφών ε, στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Έχουμε εννέα πολύ καλά μοντούλ που χρησιμοποιούμε και που ε, έχουν σχεδιαστεί και ιδιαίτερα για περιβαλλοντικά θέματα. Άρα, δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χρησιμοποιεί όλες αυτές τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν στα λιμάνια ε, και ελέγχουμε επίσης και την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Θεωρούμε ότι είμαστε βασικός πάροχος του ε, ελέγχου των ε, καυσίμων, συγκεντρώνουμε δεδομένα. Ε, κάθε ημέρα παίρνουμε πάνω από 16 εκατομμύρια μηνύματα από διάφορα σκάφη. Προσφέρουμε την επιτήρηση μέσα από τον γεωγραφικό ενταπισμό και έντεκτο Έχουμε 11.200 εικόνες που, δίδονται, που δόθηκαν εφέτος ε, στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Και χάρη των εργαλείων που έχουμε για να ανταποκριθούμε στη ρήπανση, μπορέσαμε να αξιολογήσουμε στα κράτη-μέλη όλες τις εικόνες που υπήρξαν σχετικά με τη ρήπανση. Τους τελευταίους μήνες κινητοποιήσαμε τα σκάφη μας ε, σε ατυχήματα που έλαβαν χώρα σε διάφορα μέρη του κόσμου. Επιπλέον, Επιπλέον ε, κατορθώσαμε να εκτελέσουμε 10 επιχειρήσεις κάθε χρόνο. Χρησιμοποιούμε και drone για να συμπληρώνουμε την ε, επιτήρησή μας. Ε, έχουμε 7 άρπασης ε, τα οποία αναπτύσσαμε το 2019 για τον ε, γενικότερο έλεγχο, για τον έλεγχο των εκπομπών και επίσης και για να ελέγχουμε περιπτώσεις ρήπανσης ε, λόγω πετρελοκυλίδας. Τώρα, όσον αφορά τη στρατηγική μας, πριν από ένα χρόνο προσχώρησα στην ΕΜΣΑ και το πρώτο μου καθήκον ήταν να αποκτήσουμε ένα νέο πολιτέ στρατηγικό πλαίσιο για, τη, για το φορέα μας. Αυτό το έπραξα μέσα από μια διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τα κράτη-μέλη, με τους αρμόδιους βιομηχανικούς κύκλους, με εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και με το Διοικητικό μας Συμβούλιο. Ως αποτέλεσμα αυτού έχουμε πλέον ένα φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό πρόγραμμα το οποίο αναγνωρίζει την ΕΜΣΑ ως ένα οργανισμό που βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος ε, στην τεχνολογική ανάπτυξη και ε, ως ένα πρότυπο αριστείας ε, θέματα θαλάσσιων μεταφορών. Η πενταετή μα στρατηγική βασίζεται σε πέντε πυλώνε ή πέντε S που τα λέμε από τα αγγλικά, τα αρχικά, τη σταθερότητα, τη απλούστευση, τη επιτήρηση. Για κάθε ένα λοιπόν από αυτού του πέντε στρατηγικού τομεί έχουμε καθορίσει και στρατηγικέ προτεραιότητε, όπω επίση και στρατηγικού στόχου. Και παράλληλα έχουμε καθορίσει το πώ ακριβώ θα είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτού του τομεί. Και γι' αυτό το λόγο ορίζουμε την, ε, τον ΕΜΣΑ ως ένα πάροχο υψηλής, ε, παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Βασική μας ε, εταίρη είναι βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και αυτοί από τη σειρά τους μπορούν να εφαρμόζουν και να εκτελούν τις επιχειρήσεις τους όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Θέλουμε να είμαστε αξιόπιστος εταίρος. Ο ΕΜΣΑ θα ντύνει τη συνεργασία με άλλους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρχει και περισσότερη προσθέμενη αξία για τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Εφόσον δεν μου μένει πολύς χρόνος, ε, θα μιλήσω ταχύτατα ε, θα σας παρουσιάσω τους πέντε πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι η ε, βιωσιμότητα. Στη βιωσιμότητα το πρώτο S, ε, Sustainability, αυτός είναι ο πρώτος μας πυλώνας για να στηρίξουμε το ευρωπαϊκό Green Deal και αυτό εξελίσσοντας περαιτέρω όχι μόνο τις γνώσεις μας αλλά και τα επιχειρησιακά μας καθήκοντα όσον αφορά τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα αλλά και όσον αφορά την αποκαλούμενη παραδοσία παραδοσιακή ρήπανση όπου ε, εξελίσσουμε τις δυνατότητές μας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε ενδεχόμενο ρήπανσης. Αυτά, ε, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε επανειλημμένα επισκέψεις ε, σε διάφορα, διάφορες χώρες όπου ε, θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τα εργαλεία μας. Το δεύτερο πυλώνας είναι η ασφάλεια, safety στα αγγλικά, είναι ο βασικός μας πυλώνας γιατί είμαστε οργανισμός ασφάλειας και έτσι λοιπόν έχουμε καθορίσει και έχουμε εντοπίσει ε, τα σκάφη που είναι επικίνδυνα. Είναι πολύ μεγάλα σκάφη, container και πολύ μεγάλα επιβατικά σκάφη και αλληλευτικά σκάφη, αλλά και εκείνα ε, τα οποία δεν εντάσσονται στο συμβατικό μέγεθος. Αυτές θα είναι οι προτεραιότητές μας κατά τα επόμενα πέντε έτη. Βεβαίως ε, τα μαζικά σκάφη, τα αυτόνομα σκάφη και αυτά θα πρέπει να εξεταστούν από το πρίσμα της ασφάλειας, της ε, επικοινωνίας ε, και της ζωής σε ένα ευρυδικό περιβάλλον. Θα πρέπει όμως να εξεταστούν και κάτω από το πρίσμα του ορισμού των υπηρεσιών που προσφέρει η ΕΜΣΑ. Πώς αυτά θα ενταχθούν στο νέο περιβάλλον. Στο θέμα της ασφάλειας νομίζω πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου τα βασικά στοιχεία της ασφάλειας που είναι οι άνθρωποι. Ε, έχουμε στα σκάφη ιδιαίτερα εκπαιδευμένο προσωπικό Έχουμε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όλο και περισσότερο αυτοματοποιημένα σκάφη και γι' αυτό θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και την κοινωνική διάμετρο και το θέμα της εκπαίδευσης ε, των της νέας γενιάς. Να έχει κίνητρα η νέα γενιά να κάνει αυτή τη δουλειά. Ε, θεωρούμε ότι αν ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, ε, εκεί η ΕΜΣΑ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για να είμαστε επιτυχημένοι. Βλέπετε εδώ το επόμενο που και αυτό έχει σχέση με την ασφάλεια, το ρόλο που μπορούμε να παίξουμε για να διασφαλίσουμε τον ευρωπαϊκό στόλο και πέρα από γεωγραφικές ε, ευρωπαϊκές οριζόμενες περιοχές. Εδώ μιλάμε για τρομοκρατία, για πειρατεία, για ενοπλές επιθέσεις. Ε, ο ΕΜΖΑ είναι ο βασικός φορέας ε, και μπορούμε να προσφέρουμε ε, τη θέμενη αξία. Η κυβερνοασφάλεια αυτή είναι σημαντική, οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές και λαμβάνουμε υπόψη μας και την κυβερνοασφάλεια. Επιτήρηση, έλεγχος, όπως σας είπα, ε, βρισκόμαστε στο κέντρο της θαλάσσης εικόνας και προσφέρουμε συνεχώς ε, στις διάφορες χώρες αλλά και στους αρμόδιους φορείς, υπηρεσίες γιατί αυξάνονται συνεχώς οι θαλάσσιες μεταφορές. Εμείς λοιπόν χρησιμοποιούμε την τεχνολογία που υπάρχει για να μπορέσουμε να ε, ενσωματώσουμε την τεχνογνωσία και τις πληροφορίες που λαμβάνουμε. Και ε, έτσι ε, θέλουμε και εμείς να εξετάσουμε το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε σε επιχειρήσεις διάσωσης χρησιμοποιώντας τις γνώσεις μας τις πληροφορίες που παίρνουμε από διάφορες πηγές. Όπως σας είπα, πρόσφατα παίρνουμε πληροφορίες χρησιμοποιώντας και drone, αλλά όλο και περισσότερο ελέγχουμε το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσουμε να προβλέψουμε και ή δυνατόν και να αποτρέψουμε ατυχήματα στη θάλασσα. Ένας από τους βασικούς πυλώνες ε, για μας είναι προφανώς η απλούστευση. Η ανταγωνιστικότητα της ε, ενωσιακής ε, ναυσιπλοείας βεβαίως και εξαρτάται και από τη μείωση του διοικητικού αχθούς και από τη δημιουργία μιας ενιαίας μόνο ευθυντικής ε, θηρίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω σε αυτό συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιστεύουμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στη μείωση του διοικητικού αχθού στον τομέα της ναυτιλίας. Αυτό θα έχει θετικές προεκτάσεις και στο ευρύτερο θαλάσσιο περιβάλλον γιατί θα περιστεί και ο χρόνος που δαπανούν τα σκάφη στα λιμάνια. Ως εκ τούτου θέλουμε ο έμσα φορέας μας να συμμετέχει στην ευρύτερη επιμελητιακή αλυσίδα. Ε, ξέρω ότι έχω ξεπεράσει το χρόνο που έχετε προβλέψει για μένα. Θα ήθελα μόνο να πω κάτι τελευταίο και να το υπογραμμίσω. Ξέρετε, εμείς χρησιμοποιούμε κατά κόρον την τεχνολογία, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι το ουσιαστικό μας κεφάλαιο είναι το προσωπικό μας. Έχουμε 270 ε, προσοντούχους ε, υπαλλήλους με πάρα πολλά προσόντα και με τέτοιο κεφάλαιο μπορεί κανείς να προβληθεί δίνοντας το καλό παράδειγμα. Είμαστε εκείνος ο Φαρέας που έχει και στην καρδιά του και στην εντολή του το πρασίνισμα, το περιβάλλον. Ε, έτσι λοιπόν πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα όπως σας είπα και για το λόγο αυτό έχουμε ξεκινήσει ένα ε, πρόγραμμα το που λέγεται πρασίνισμα του ΕΜΣΑ και αυτό σημαίνει ότι εφαρμόζουμε ένα δικό μας σύστημα με διάφορα μέτρα ε, και με τον τρόπο αυτό ε, θα δείξουμε τον δρόμο, θα δώσουμε το καλό παράδειγμα ε, με άλλα λόγια, ε, δεν χρησιμοποιούμε πλαστικές ε, ύλες, ηλεκτρική ενέργεια, κατά 100% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε σε βιωσιμότητα στους δημόσιους διαγωνισμούς και στις εγκαταστάσεις μας χρησιμοποιούμε ηλεκτρικά οχήματα. Ε, εν ολίγης προσπαθούμε και να κάνουμε και άλλα, παραδείγματος χάρη να καθαρίσουμε τις ε, παραλίες γύρω από την ε, Λισαβόνα. Γύρω από την Λισαβόνα. Θέλω λοιπόν να μας επισκεφτείτε και ή δυνατόν να συνεργαστείτε μαζί μας στο να ε, πρασινίσουμε τον ΕΜΣΑ ε, που είναι ένας εμβληματικός αποκεντρωμένος οργανισμός τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπάμαι που μακρηγόρησα, ελπίζω να ήμουν ε, κατανοητή. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Αρχίζει η συζήτηση, διότι όπως είπατε υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις στον τομέα της ναυτιλίας και των θαλασσίων μεταφορών. Όπως είπατε, το, η κλιματική αλλαγή είναι επίσης για σας ένα θέμα σημαντικό. Πώς θα συμμετάσχετε στο περίφημο πρασίνισμα, το Green Deal της Κομισιόν. 55% μισθ. Πώς θα μπορέσετε εσείς να ε, ενεργήσετε συγκεκριμένα ώστε να αποδεσμευτείτε από τον άνθρακα, να κάνετε πιο πράσινα τον τομέα της δικής σας ε, θητείας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας. Θα δώσω το λόγο, αυτή ήταν μια γενική ερώτηση, δίνω το λόγο και σε άλλους συναδέλφους. Εκ μέρους του ΕΛ και δύο λεπτά κυρία Τέλλερ. Σας ευχαριστούμε κυρία Κώστελακ για την εμπεριστατωμένη ανάλυση του οργανισμού σας. Συγχαρητήρια που μας, για την παρουσίασή σας. Είμαι από την Αυστρία. Για μας το νερό και κυρίως το νερό της θάλασσας δεν είναι η ειδικότητά μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αναγνωρίζω πόσο προστιθέμενη αξία παρέχει ο οργανισμός σας. Σας ευχαριστούμε, λοιπόν. Έχω μία ερώτηση που αφορά την εποπτεία και τα μέσα αυτοματοποιημένης εποπτείας για να μπορέσετε να ανοιχτεύσετε ανώμαλες συμπεριφορές και τους αλγορίθμους που χρησιμοποιείτε που είναι ένα ισχυρό αναλυτικό εργαλείο. Είπατε επίσης ότι χρησιμοποιείτε τα ντρόν και διαστημικούς σταθμούς που εκπέμπουν για να μπορέσετε να ξέρετε τι ακριβώς γίνεται για την εποπτεία. Πώς ένα σκάφος μπορεί να πλέει στην ε, Μεσόγειο χωρίς να ανοιχνεύεται από όλα αυτά τα μέσα. Τι πρέπει να αλλάξει και τι δυνατότητες περαιτέρω εποπτείας χρειάζεστε για να φέρετε σε πέρα στην αποστολή σας. Ευχαριστώ. Κύριος Δάνιλσον. Λιγότερο Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και για την παρουσίαση. Θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω σου ειδικά. Η ΕΜΣΑ στην ιστοσελίδα της αναφέρεται στο γεγονός ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για ατυχήματα επειδή υπάρχει ε, περισσότερη κυκλοφορία. Ε, αυτό βεβαίως επηρεάζει και το περιβάλλον, επηρεάζει και τους εργαζόμενους στα πλοία. Μας περιγράψατε σήμερα πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους αυτούς μέσω της τεχνολογίας, μέσω και κανονισμών βεβαίως και κανόνων. Ε, το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξή. Εσεί θεωρείτε ότι εμεί ω νομοθέτε πρέπει να θέσουμε ω προτεραιότητα να έχουμε έναν ασφαλή ε, χώρο εργασίας για τους εργαζόμενους. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό, πώς μπορούμε επίσης να μειώσουμε τον αντίκτυπο αυτής της αύξησης της ε, κυκλοφορίας στο περιβάλλον κύριος Δίας δεν θέλει το λόγο. Δεν θέλετε το λόγο, κύριε Μπαθαντίας. Δεν θέλετε. Εντάξει. Ο κύριος Κοφ έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ και για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, κυρία Κώστελατς. Ε, στην παρουσίασή σας αναφερθήκατε ε, σε πάνω από 3.000 ατυχήματα το χρόνο. θα ήθελα να αναφερθώ τώρα εγώ στην απώλεια ανθρώπινων ζωών. Πού έχουμε απώλεια ζωής. Ποιες είναι οι τάσεις σε ό,τι αφορά τα θανατηφόρα ατυχήματα στα ευρωπαϊκά ύδατα και λίγο πιο συγκεκριμένα τώρα σε ό,τι αφορά τον τραγικό αριθμό απώλεια ζώων στη Μεσόγειο. Για τους ανθρώπους, ε, από τους ανθρώπους που προσπαθούν ε, να φτάσουν στην Ευρώπη ε, με διάφορα μέσα τα οποία είναι εντελώς ακατάλληλα. έχετε κάποιο σχόλιο εσείς για τον αριθμό των πνιγμένων αυτών ανθρώπων και κάτι ακόμα σε σχέση με τους, ε, ε τις αρχές φάρων ε, της Ευρώπης και τους νέους ρόλους που έχουν αναλάβει ε, πώς η δική σας υπηρεσία ε, συνεργάζεται με τις διάφορες ε, υπηρεσίες φάρων την Ευρώπη. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε πρώτα για τις απώλειες ζωής, γενικότερα ποιες είναι οι τάσεις και ειδικότερα για τη Μεσόγειο και τους πρόσφυγες και, το, και δεύτερον οι σχέση σας με τις διάφορες αρχές ε, φάρων. Ε, ναι, θα δώσω τώρα το λόγο στο όνομα της κυρίας Ρινιού, την κυρία Νάτιγκαλ. Ε, πρώτα δίνουμε το λόγο στους συντονιστές, Εντίτ, έτσι. Είναι η αρχηγή, ας πούμε, του κόμματος και μετά στους βουλευτές, εντάξει. Έτσι κύριε Ρικέ, καλό είναι να ενημερώνουμε τους ανθρώπους. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την παρουσίαση. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο ε, στο εργαλείο Net, Δημιουργήθηκε για να μπορούμε να αντιδρούμε πιο γρήγορα όταν έχουμε ατυχήματα, δυστυχήματα, ε, επικίνδυνες καταστάσεις στη θάλασσα σε αυτά τα συστήματα παρακολούθησης ε, συλλέγονται στοιχεία και αποθηκεύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό είναι εξαιρετικά θετικό, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Αυτά τα δεδομένα προέρχονται από τις λιμενικές αρχές, από τις, τους ε, και μπορούμε να έχουμε τις πληροφορίες αυτές. Δυστυχώς όμως ε, στον κλάδο αυτών υπάρχουν ορισμένες περιπλοκές ε, αχρίαστες διαδικασίες προβληματικές Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε αυτό και ποιος είναι ο ρόλος που μπορεί να παίξει η ΕΣΜΑ. Διότι ε, όταν μιλάμε για την ασφάλεια στη θάλασσα, ε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα της αξιοπιστίας ε, και της ε, ε, απλότητας, της ταχύτητας με την οποία μπορούμε να κινηθούμε. Η κυρία Κουντουρά έχει το λόγο. Όχι, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, ο κύριος Ζήλε. Ναι. Ε, Μάλιστα. Ε, δεν με... Ε, δεν με γι' αυτό, έτσι. Δεν σας πειράζει. Ε, θα μας συγχωρέσετε. Ναι, απλώς ξέρω την μου. Να πάρω το λόγο. Ευχαριστώ την κυρία Κώστελα για την παρουσίαση. Ήμουν στη Λισαβόνα, στην έμψα πριν βέβαια στη δική εποχή. Ήταν πραγματικά ε, προφανές ότι υπήρχαν μεγάλες τεχνικές δυνατότητες, υπήρχαν και δυσκολίες όμως στη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών της Ένωσης για τις ζητήματα ασφάλειας, Frontex, EMSA, ε, διότι ορισμένε φορές ε, κάποιοι κατεβάζουν τα συστήματα πληροφοριών, εσείς μπορούσατε να δώσετε πληροφορία στην Frontex, στην για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Τι γίνεται όμως, ε, ε, υπάρχει κάποια βελτίωση, διότι η μεταφορά των ε, μεταναστών οδηγεί στις τραγωδίες. Έχετε καλή συνεργασία με την Frontex για τα ζητήματα ασφάλειας. Ευχαριστώ τον κύριο Ρόμπερτ Τζίλε. Κυρία Κουντουρά έχει το λόγο, παρακαλώ. Πρόεδρε, ε, θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας και είναι ιδιαίτερα μάλιστα μεγάλη χαρά που σας έχουμε κοντά μας μια γυναίκα σε θέση ευθύνη σε έναν κατά τα άλλα ανδροκρατούμενο κλάδο. Ο οργανισμός του οποίου ηγείστε έχει θέσει πολύ φιλόδοξους στόχους για την επόμενη πενταετία και θα ήθελα να σταθώ στο θέμα της βιωσιμότητας μιας και είναι η οριζόντια προτεραιότητά μας για τα επόμενα χρόνια. Σωστά το εντοπίζετε και εσείς στη στρατηγική σας ε, και θα ήθελα να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένοι σχετικά με τα εργαλεία που σκοπεύετε να αναπτύξετε τα επόμενα πέντε χρόνια και ειδικά για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης αλλά και της θαλάσσιας ρήπανσης. Αναφέρεστε σε αυτά τα προβλήματα αλλά δεν αναπτύξατε συγκεκριμένες προτάσεις. Είναι σημαντικό ε, το κομμάτι των δραστηριοτήτων σας και αφορά τόσο την πρόληψη όσο και την αντιμετώπιση της ρήπανσης από πλοία είτε λόγω ατυχημάτων είτε λόγω παράνομων ε, ενεργειών. Και στο επίπεδο της πρόληψης υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης καθώς από το 2011 ως το 2017 είχαμε στην Ευρώπη 603 ναυάγια και 683 θανάτους. Πώς σκοπεύετε να βελτιώσετε αυτά τα απαράδεκτα στατιστικά και τέλος, στο, τέλος, στο σκέλος της αντιμετώπισης ατυχημάτων από την εμπειρία σας πώς θεωρείτε ότι μπορεί να βελτιωθεί η συνεργασία σας με τα κράτη μέλη σε θεσμικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για το ερώτημα. Κυρία Μοντέρο, έχετε το λόγο. Παρακαλώ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την προσκεκλημένη μας για την παρουσίαση που έκανε και όντως πρέπει να πω ότι αναγνωρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο κάνετε. Το έργο σας το αναγνωρίζουν τα κράτη-μέλη και εμείς. Και όλοι. Όσον αφορά την ψηφιοποίηση, την ασφάλεια και την καταπολέμηση των κλιματικών προβλημάτων. Ξέρουμε ότι πρέπει να έχουμε ε, στόλους πιο καθαρούς, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι, ποια είναι τα προβλήματα που αφορούν επίσης τη μισθή της και όλα τα θέματα τα οποία είναι της αρμοδιότητας της δικής μας και της δικής μας στον τομέα της ε, θαλάσσιων μεταφορών. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα που χρησιμοποιείται, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να μειώσουμε ποσοστό του του άνθρωπου, τις εκπομπές και πώς θα μπορέσουμε να έχουμε την κατάλληλη νομοθεσία πλαίσιο σχετικά με αυτό το θέμα στα κράτη-μέλη. Σε σχέση τώρα με αυτό το οποίο είπαμε και κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα ψήφισμα για την COP25 και για τις θαλάσσιες μεταφορές. Πώς βλέπετε ότι είναι έτοιμος ο τομέας των θαλασσίων μεταφορών ε, ε, φτάσει τους στόχους αυτούς. Είναι προετοιμασμένος. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με πιο καθαρά καύσιμα, με μεταβατικής περίοδου καύσιμα, το LNG. Πώς το βλέπετε όλο αυτό το θέμα σε σχέση με την αύξηση χρησιμοποίηση αυτού του καυσίμου. Επίσης, τι έχετε να μας πείτε για τον τρόπο διαχείρισης διαφόρων θεμάτων στα διάφορα λιμάνια της Ευρώπης εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ποιο τρόπο μπορούμε να υποστηρίξουμε περισσότερο ή να βοηθήσουμε την ναυτιλία για την μείωση των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακος και πώς μπορούμε επίσης να συνεργαστούμε και με εσάς και με την ΆΙΜΟ. Ευχαριστώ. Κύριος Λιμπεράσκη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όντως ε, αυτά που είπατε κύριε Κώσταλατς είναι ε, αλήθεια. Οι ευρωπαϊκές μεταφορές είναι ε, στα χέρια γυναικών. Επίτροπος, εσείς εδώ στην Επιτροπή μας. Αντιμετωπίζουμε όμως ένα ζήτημα. Ήμουν και εγώ στην ψηφοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου θεωρούν ότι η ΕΜΣΑ δεν ενδιαφέρεται σε ό,τι αφορά το, τα γιότ. Ήμουν στην Ένωση την Ευρωπαϊκή για τον γιότ, έτσι. Μιλάμε για πάνω από 8,5 μέτρα, έτσι. Έχουμε στατιστικά στοιχεία τα οποία ε, δεν είναι συμβατά. Επίσης υπάρχει το θέμα της, του παροπλισμού των πλοίων επειδή είναι, μπορεί να είναι μικρά τα πλοία αυτά, αλλά είναι εκατομμύρια στα ύδατα της Ένωσης. Είναι ένα καλό μοντέλο τουρισμού, είναι ένα καλό μοντέλο διαχείρισης των υδάτων γενικότερα. Τώρα, ένα άλλο ερώτημα. Υπάρχει ένα θέμα ασφάλειας όχι μόνο για τα πλοία, αλλά και για τους ανθρώπους ένας ε, ε, πλοίαρχος ε, Πολωνός ανέφερε στη Λατινική Αμερική ότι είχε την υποψία ότι ένα κοντέινερ περιείχε προϊόν λαθρεμπορίου. Και ήταν αλήθεια. Αλλά έχει συλληφθεί ο άνθρωπος αυτός. Ο, ο άνθρωπος το ανέφερε και κανείς δεν μπορεί να το βοηθήσει. Τι γίνεται για αυτές τις περιπτώσεις όταν μιλάμε για την ασφάλεια. Έτσι, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας, αλλά ασφάλεια και των ανθρώπων. Και τέλος, υπάρχουν στοιχεία για την ποιότητα του προσωπικού, του πληρώματος των πλοίων. Πριν από μερικά χρόνια στο Κοινοβούλιο είχαμε εγκρίνει ε, κάποια, ένα κανονισμό μάλλον για, τα, ε, για τις ποιοτικές προδιαγραφές ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση, παρουσίασή σας, διότι μάθαμε πολλά. Ευχαριστώ κύριε Λιμπεράτσκι. Πριν δώσω το λόγο ε, στην, συνάδελφο, ε, έχουμε εδώ και κάποιον παλιό που δεν θέλει να φύγει από Επιτροπή μεταφορών, ε, ο κύριος Βιμ Βαντενκάμπ, ο οποίος είναι ξανά στην Επιτροπή Μεταφορών, εκ νέου. Καλώς ήρθατε. Βιμ, ελπίζω να είστε καλά. Ναι, βεβαίως, είμαι ένας πλούσιος συνταξιούχος, πολλά λεφτά, πολύς χρόνος και νιώθω πολύ καλά. Βέβαια, εντάξει, έχω και μια νοσταλγία. Σας ευχαριστώ. Πάντως είστε πάντα καλοδεχόμενοι στην Επιτροπή μας. Ε, ε, αλλά να προσέχετε τι καταναλώνετε, διότι η κατανάλωση κάνει κακό στον πλανήτη. Με τα χρήματά σας εννοώ. κυρία Μπιλμπάου έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλες και όλους. Ε, να καλωσορίσω και την ε, προσκεκλημένη σήμερα. Πρέπει να θυμίσουμε ότι η ΕΜΣΑ, όπως και άλλα πολλά ευρωπαϊκά project, προέρχονται από δύο μεγάλα ατυχήματα, το ΕΡΙΚΑ και το Prestige και βεβαίως έχουμε αναθεωρήσει ε, την, ε, τις αρμοδιότητες της ΕΜΣΑ, τις έχουμε ενισχύσει πάντα συναντώντας αντίσταση, όμως ε, φάνηκε για άλλη μια φορά ότι είναι περισσότερο σημαντική και απαραίτητη από ποτέ αυτή η υπηρεσία και οι αρμοδιότητες της. Πέρα από τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε, θα ήθελα να σας συγχαρώ βεβαίως για το θέμα ε, της ισότητας μεταξύ των δύο φίλων ε, που μας, μας απασχολεί ε, και βλέπω ότι την κάνατε πραγματικότητα. Ε, η συνεργασία σας, ε, της υπηρεσίας σας μάλλον με την ε, Επιτροπή Ελέγχου της Αλίας, πώς πάει. Εγώ είμαι και στις δύο επιτροπές, και την Επιτροπή Αλίας δηλαδή και αυτήν. Θα ήθελα να ξέρω αν θεωρείτε ότι υπάρχει, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης Πρώτον, με την, τον, με την ε, Επιτροπή Ελέγχου της Αλίας και σε ό,τι αφορά τον, την υπηρεσία ελέγχου των θαλάσσιων μεταφορών για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Ε, ξέρετε ότι βρήκαμε ένα υποβρύχιο με ποσότητες ε, ναρκωτικών ε, πραγματικά κλίμακα επιστημονικής φαντασίας, κοντά στη Γαλλικία. Ε, θεωρείτε ότι έχετε τους απαραίτητους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για να μπορείτε να ανταποκριθείτε ε, σε όλα αυτά τα πράγματα που απαιτούμε από εσάς αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ την κυρία η Κυρία Ντεπαρνέ, καλώς ήρθατε, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Κώστελατς, χαίρομαι που σας βλέπω εδώ. Όπως είπε και η Πρόεδρος, πλέον ε, πάμε μαζί προ ένα κόσμο χωρί ορικά καύσιμα, ελπίζουμε να πηγαίνουμε προ τη κατεύθυνση. Τώρα δεν ξέρω αν η ΕΜΣΑ έχει απόψει για τον κίνδυνο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και των σχετικών ε, εγκαταστάσεων στα ύδατα τη Ένωση. Θα είχε νόημα να υποστρίξουμε περαιτέρω την οργάνωση αυτή ε, και να για, να πάρθουν μέτρα ε, εφόσον υπάρχουν περαιτέρω κίνδυνοι λόγω αυτών των πλατφορμών. Και θα ήθελα να ξέρω όπως είπε η κυρία Νότιγκαλ σα ρώτησε, ε, σε σχέση με το net ε, υπάρχει χρηματοδότηση για, την, για τα προγράμματα ψηφιοποίηση, παραδείγματο χάρη, ε, σε σχέση με τι πλατφόρμε αυτέ. Μάλιστα. Ευχαριστώ την κυρία Ντεπαρνέ. Ο κύριος Νοβάκοφ έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Κώστελατς, ε, θα ακολουθήσω ε, το παράδειγμα της Μπαρατάλτερ. Προέρχομαι και εγώ από μια ορεινή περιοχή, έτσι, οπότε ούτε εμένα η θάλασσα είναι ο φυσικός μου χώρος. Είμαι σε μια χώρα όμως που έχει και βουνά και θάλασσα. Όλο και πιο πολλά ευρωπαϊκά πλοία έχουν μη ευρωπαϊκή σημαία για διάφορους λόγους κυρίως επειδή από οικονομικής πλευράς είναι πιο συμφέρον ε, να επιλέγει κανείς άλλη σημαία από οπουδήποτε στον κόσμο αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται λόγω χαμηλότερων οικολογικών προδιαγραφών όμως. Ε, εσείς ε, πιστεύετε ότι υπάρχει δυνατότητα να προσελκύσουμε αυτούς τους πλειοκτήτες ε, να εγγράψουν τα πλοία τους ε, σε ευρωπαϊκά μητρώα με ευρωπαϊκή σημαία να πληρώνουν και φόρους εδώ αντί να χρησιμοποιούν ε, αυτές τις νομικές πρακτικές που τους επιτρέπουν να εγγράφονται στο εξωτερικό. Κύριε Ρικέ, έχετε το λόγο παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να και την κυρία Μάρκοβιτς Κώστελετς για τα, την παρουσίασή της δύο ερωτήματα. Ε, Βεβαίω εδώ έχω μια ερώτηση που αξίζει 25 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το λέω αυτό γιατί η Ευρώπη έχει και υπερπόντια εδάφη και εκεί υπάρχουν τεράστια, ε, τεράστιες εκτάσεις ε, θαλάσσιες. Τι κάνετε για αυτές τις περιοχές, ε, τι σχέσεις έχετε μαζί τους, ε, Υπάρχει κάποιο σχέδιο που να σας επιτρέπει να, είστε πιο, να είναι πιο έντονη η παρουσία σας στις περιοχές αυτές όπου τα συμφέροντα τα ευρωπαϊκά είναι τεράστια. Ε, και τώρα σε ό,τι αφορά το περιβαλλοντικό σας, ε, τους περιβαλλοντικούς σας στόχους, ε, εσάς έως τώρα εσείς ασχολείστε κυρίως με την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ατυχημάτων, δηλαδή γεγονότων μη επιθυμητών. Ε, τώρα θα έχουμε και έναν επίτροπο για τους ωκεανούς όμως στα πλαίσια του Green Deal. Η κατάσταση λοιπόν σε ό,τι αφορά τους ωκεανούς και την ποιότητα των ωκεανών θα μας απασχολήσει. Ποιες είναι οι σχέσεις σας με τις άλλες ε, γενικές διευθύνσεις της Κομισιόν ε, αυτή που θα δημιουργηθεί παραδείγματος χάρη τώρα για, αυτή, για τους ωκεανούς και κατά πόσο έχετε σχέσεις με κάποια επιστημονικά Ινστιτούτα ευρωπαϊκά που είναι επιφορτισμένα με την παρακολούθηση ε, της κατάστασης των ωκεανών. Μάλιστα ευχαριστώ τον κύριο Ρικέ. Είχα και εγώ ένα τελευταίο ερώτημα να θέσω. Μιλήσαμε ε, για τα απορρίμματα νωρίτερα. Τα απόβλητα ιδιαίτερα ε, στον τομέα των το θαλάσσιο είναι όλο και πιο έντονο αυτό. Ε, έχετε δίκιο και εσείς κύριε Τι θα κάνετε έτσι ώστε και ο τομέας θαλάσσιων μεταφορών να μπει στην οικολογική μετάβαση. Και ένα τελευταίο ερώτημα που είναι πολύ σημαντικό θεωρώ και που νομίζω δεν το προσεγγίζουμε απαρκώς. Το θέμα της ρήπανσης της ατμόσφαιρας διότι οι θαλάσσιες μεταφορές επηρεάζουν την ρήπανση της ατμόσφαιρας και αν επιστρέφω στο θέμα της Μεσογείου εδώ βλέπουμε ε, αυτά τα πλοία που εκπέμπουν θείο, διοξείδιο του άνθρακα ε, σωματίδια και όλες αυτές οι πόλεις που ε, φιλοξενούν αυτά τα πλοία τα μεγάλα πλοία, ε, ασφικτιούν. Θα μας βοηθήσετε λοιπόν έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτές τις παρήφημες ζώνες χαμηλών εκπομπών. Οδηγίες όπως η οδηγία για το θείο να μπορέσουν να ενισχυθούν. Ε, να δούμε τι θα γίνει με τα καύσιμα αυτών των πλοίων. Δεν μπορούμε πια να αναπνεύσουμε, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο ε, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάναμε στο βορρά, έτσι. Ε, στη Βόρεια Θάλασσα, όπου έχουμε αυτές τις ζώνες ε, χαμηλών εκπομπών. Θα είναι νομίζω μια από τις μεγάλες προκλήσεις της θητείας αυτής να δημιουργήσουμε αυτές τις ζώνες έτσι ώστε αυτά τα πλοία να μην πλήττουν την υγεία των κατοίκων που ζουν κοντά στα λιμάνια αυτά. Επίσης υπάρχει το θέμα του εξοπλισμού, διότι και αυτό θα μας απασχολήσει. Ε, αυτά τα πλοία που δεν έχουν βεβαίως ε, η, τέτοια βαριά καύσιμα, αλλά πώς θα τα εξοπλίσουμε καταλήλως. Ε, να δούμε ποιο είναι, να δούμε και το θέμα των, του μεγέθους αυτών των πλοίων, που δεν είναι πια πλοία, έτσι είναι κινούμενα νησιά. Είναι τεράστια. Είχαμε, αυτή την εικόνα στη Βενετία και είναι το τεράστιο πλοίο που φτάνει. Ε, δεν γίνεται. Ε, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για την ασφάλεια, όταν μιλάμε για τις εκπομπές. Ε, δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια πλοία στο μέλλον. Ξέρω ότι είναι πολλά τα ερωτήματα. Θα έχετε και λίγο χρόνο. Κάτι παραπάνω από 6 λεπτά θα σας δώσω ε, για να απαντήσετε. Έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Thank you, Madam. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους ε, για τα σχόλιά σας και τις ε, ερωτήσεις και θα προσπαθήσω κάπως να ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις. Θα απαντήσω στα βασικά θέματα που θέσατε. Πρώτα απ' όλα υπάρχει προφανώς το τι ακριβώς κάνουμε σε θέματα περιβάλλοντος και ναυτιλίας ε, ετέθησαν αρκετά θέματα. Θα θίξω το θέμα της κλιματικής αλλαγής, το Green Deal, την ε, ρήπανση, ρήπανση από τα σκάφια αλλά και από τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Ο ΕΜΣΑ, ο οργανισμός μας, αναμφισβήτητα έχει ένα ρόλο να παίξει, δηλαδή να βοηθάει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ε, κυρίως ε, όσον αφορά στην ε, συγκεκριμενοποίηση όλων των στοιχείων της, του Πράσινου Συμφώνου. Δηλαδή η νομοθεσία που πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή. Ε, ο ΕΜΣΑ καλείται να στηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη στο στοιχείο της ε, τεχνογνωσίας. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Βελτιώνουμε συνεχώ τις γνώσεις μας για να μπορέσουμε να επιτελέσουμε το καθήκον μας. Παράλληλα, συμμετέχουμε στον ε, διεθνή διάλογο ε, προβάλλοντας τα ευρωπαϊκά επιχειρήματα σε διεθνές ε, πλαίσιο. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ναυτιλία εξορισμού είναι διεθνής και αυτό που έχει σημασία είναι να επιτυγχάνουμε συνένεση και λύση κυρίως για τα περιβαλλοντικά θέματα σε παγκόσμια βήματα. Εδώ λοιπόν είναι σημαντικό η Ευρώπη να μιλάει με μία φωνή. Ο ΕΜΣΑ έχει τη δυνατότητα να διευκολύνει το διάλογο και τις διαπραγματεύσεις. Πιο συγκεκριμένα, επειδή πρόκειται για ένα πολύ περίπλοκο θέμα, δεν πρόκειται μόνο για την ναυτιλία η οποία πρέπει να αλλάξει. Είναι και το θέμα των λιμανιών γιατί αναφέρεται το θέμα των εναλλακτικών καυσίμων ως μία από τις λύσεις ε, για να ελέγχονται οι εκπομπές ε, τόσο διοξιδίου όσο του άνθρακα όσο και του αζότου. Ε, ως εκ τούτου καλούμεθα να μετακινηθούμε από τα παραδοσιακά ορυκτά κάψιμα μέσα από το υγροποιημένο φυσικό αέριο ε, στην αλλακτική λύση που είναι τα μη ορυκτά κάψιμα. Άρα δηλαδή όλοι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Και εκείνο το οποίο κάναμε είναι να δώσουμε οδηγίες ε, για την χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Αυτό ήταν ε, ένα από τα σημαντικότερα έγγραφά μας ε, στην εισήγησή μας. Βοηθάμε και τις δύο πλευρές της ε, βιομηχανίας έτσι ώστε να υπάρχει σωστή λειτουργία ε, όσον αφορά τη χρήση των σκαφών. Και το ίδιο θα κάνουμε και για άλλα εναλλακτικά κάψιμα. Αυτή είναι ε, η απάντηση και σε μία από τις ερωτήσεις. Δηλαδή, συνεργαζόμαστε σε διάφορα επιστημονικά προγράμματα, ε, κυρίως ε, σε εκείνα που χρησιμοποιούνται από την ΕΝΕΑ και συμμετέχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο των οργανισμών που εφαρμόζουν τέτοια προγράμματα. Αποτέλεσμα ότι υπάρχουν συγκεκριμένες συνεισφορές δικές μας σε συγκεκριμένες δράσεις. Όσον αφορά τώρα στο ρόλο του φορέα μας, του ΕΜΣΑ. Βεβαίως ε, και είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος μας ε, όσον αφορά ε, την εναρμοσμένη εφαρμογή των στοιχείων. Αυτό λέγεται θέτης και αποτελείται από νέα μοντούλ. Ανέφερα στην παρέμβασή μου ότι ασχολούμαι κυρίως με θέματα εκπομπών στην ατμόσφαιρα. Δηλαδή, βοηθάμε τα κράτη-μέλη να κάνουν καλύτερους ε, ελέγχους ε, των εκπομπών. Αυτό είναι το πρόγραμμα EU Thetis, το οποίο διασφαλίζει την σωστή εφαρμογή ελέγχων σκαφών που χρησιμοποιούν ε, καύσιμα που περιέχουν θείο καύσιμα. Σχετικά πρόσφατα έχουμε αναπτύξει και ένα άλλο πρόγραμμα για να βοηθάμε στην εφαρμογή της οδηγίας MRV. Συγκεντρώνουμε πληροφορίες για εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από σκάφη και μπορώ να σας πω ότι όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν μία βάση συζητήσεων που γίνονται σε σχέση με το διοξίδιο του άνθρακα. Ε, με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο βοηθάμε τα κράτη-μέλη. Σας είπα ότι πρόσφατα ε, έχουμε συμπεριλάβει στις, ε, στο χαρτοφυλάκιό μας τις εργασίες μας και τα drones, τα μη παντρωμένα σκάφη. Χρησιμοποιούμε drones που είναι εξοπλισμένα με τα αποκαλούμενα sniffer. Τα sniffer αυτά ελέγχουν τις εκπομπές από μεμονωμένα σκάφη. Αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τα λιμάνια, γιατί με τρόπο αυτό εντοπίζονται τα σκάφη τα οποία ξεπερνούν το όριο ε, χρήσης θείου που επιτρέπεται. Τον έλεγχο των εκπομπών αζότου και άλλων ε, απαγορευμένων ιών αυτό το όριο το έχουμε εισαγάγει στη Μεσόγειο και σε άλλες περιοχές σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και με άλλους ε, και με άλλα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Μεσογείου. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα τέτοιο εργαλείο κοινό για το σύνολο της Μεσογείου. Εμείς λοιπόν διευκολύνουμε όλες αυτές τις συζητήσεις, συμμετέχουμε ενεργά στις συζητήσεις και όχι μόνο αυτό αλλά έχουμε και το πρόγραμμα ΘΕΦΑΜΕΔ, το οποίο χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με αυτό το πρόγραμμα ε, στηρίζουμε ε, τα μεσογειακά κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δυνατότητά τους να μπορούν ουσιαστικά να εφαρμόζουν στο εγγύς μέλλον, ελπίζω τουλάχιστον, ελέγχους ε, σε απαγορευμένες εκπομπές στη Μεσόγειο. Όταν πρόκειται για την πιο παραδοσιακή ρήπανση του πετρελαίου. Ξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα. Προσπαθούμε να επεκτείνουμε περαιτέρω το δικτυό μας, το χαρτοφυλόκιο που, έχουμε, ε, που έχουν ενταχθεί σκάφη, αλλά όχι μόνο σκάφη, αλλά και δύο ε, διαφορετικές ε, εργαλειοθήκες Εκεί χρησιμοποιούμε την αξιολόγηση κινδύνων. Ε, καλύπτουμε λοιπόν ε, όλη τη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης. Και πέρα από αυτό χρησιμοποιούμε και το Cleasing Net. Ε, πρόκειται ένα σύστημα γεωγραφικής παρακολούθησης που δίνει τη δυνατότητα έγκαιρα να εντοπίζουμε πετρελοκυλίδες για να αντιδρούμε με ταχύτητα. Βλέπουμε λοιπόν το πώς ε, με συγκεκριμένα μέτρα ε, μπορούμε να δράσουμε και προληπτικά γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούμε να συμβάλλουμε σημαντικά ε, στον περιορισμό παράνομων πετρελοκυλίδων γιατί η ναυτιλία και η σχετική βιομηχανία γνωρίζει πολύ καλά ότι εξακολουθεί να χρησιμοποιείται πετρέλαιο και να προκαλούνται προβλήματα. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιούμε τους πόρους μας και για πρόληψη. Όσον αφορά τώρα στους οικονομικούς πόρους που διαθέτουμε, οποτεδήποτε μπορούμε, ε, τους χρησιμοποιούμε, όπως είπα προηγουμένως, και για να προστατεύουμε την ευρωπαϊκή ναυτιλία με τον κόσμο. Χρησιμοποιούμε εργαλεία που μας επιτρέπουν να ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Έχουμε και ένα πρόγραμμα το οποίο εισαγάγαμε πρόσφατα. Είναι ένα δορυφορικό σύστημα το οποίο επιτρέπει την ε, παγκόσμια κάλυψη ελέγχων. Και εκεί, ε, όποτε το ζητούν τα κράτη-μέλη, αναπτύσσουμε και συστήματα γεωγραφικής παρακολούθησης σε απομονωμένες ε, περιοχές ή σε τρίτα εδάφη. Όσον αφορά στις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα και την COP25, ε, όπως είπα, η ενεργειακή αποδοτικότητα προβλέπει διάφορα μέτρα για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που συζητούνται σε διάφορα επίπεδα Μόλις φέτος δημοσιεύσαμε την πρώτη έκθεση που έχει σχέση με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από τα σκάφη που έχουν ευρωπαϊκή σημαία, αλλά και από σκάφη τα οποία ελιμενίζονται σε ευρωπαϊκά λιμάνια. Τα κρουαζιερόπλια αναφέρθηκαν στη στρατηγική μας, ε, για πρώτη φορά θα έλεγα, αναφέρουμε ειδικά τα σκάφη τα οποία πλέουν κάτω από, από το συμβατικό μέγεθος. Αναφέρομαι στα κρουαζιερόπλαια. Εγώ είμαι από την Κροατία και ξέρω πολύ καλά ότι αυξάνεται συνεχώς ε, αυτός ο αριθμός των ε, ε, μικρών σκαφών, των κρουαζιερόπλαιων και αυτά ε, είναι, έχουν σημασία για τη βιωσιμότητα, για το περιβάλλον, αλλά και για θέματα ασφάλειας. Στη στρατηγική μας, λοιπόν, αναφέρουμε το ρόλο που μπορούμε να διαρματίσουμε στο μέλλον, σε αυτό το τομέα, κυρίως ε, όσον αφορά ακριβώς αυτό το θέμα του χαρτοφυλακίου μας που αφορά στα κουρασγερόπλια. Η ασφάλεια η ασφάλεια παραμένει στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Το πρώτο ερώτημα είχε σχέση με τις τάσεις ε, που επικρατούν. Ποια είναι η ε, διαφανόμενη τάση για ατυχήματα σε ε, ευρωπαϊκά ύδατα. Θα έλεγα ότι είναι σταθερή. Πριν από τρία χρόνια περιορίστηκε ο αριθμός, έκτοτε παραμένει σταθερός Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε κατά 100% ικανοποιημένοι γιατί θέλουμε η τάση να εκμηδενιστεί ή αν όχι να, περιοριστεί σημαντικά, να περιοριστούν τα ατυχήματα στα ευρωπαϊκά ύδατα και από σκάφη με ευρωπαϊκή σημαία. Εδώ αναφέρομαι κυρίως στα αλλιευτικά σκάφη. Εκεί υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτιώσεων. βελτίωση στο νομοθετικό στοιχείο, στην εφαρμογή των αποφάσεων, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, θα εστιάσουμε τις ε, προσπάθειές μας στα μεγάλα σκάφη. Βέβαια αυτά είναι αρκετά δύσκολα, περίπλοκα και υπάρχουν πολλές ανησυχίες ε, σχετικά με τις δυνατότητες κένωση του σκάφου σε περίπτωση ατυχήματο. Θα εστιάσουμε όμως την προσοχή μας και στα αλλιευτικά σκάφη, όπου μεγάλο ρόλο παίζει η εκπαίδευση ε, του προσωπικού που βρίσκεται πάνω στο σκάφος ε, και αυτό αφορά και άλλους ε, και ευρύτερο προσωπικό που δεν είναι εκπαιδευμένοι ναυτεργάτες. Συνεργαζόμαστε και με άλλους φορείς Ξετάζουμε θέματα ασφάλειας. Θα γνωρίζετε φαντάζομαι ότι το 2016 ε, έληξε η δική μας η εντολή αλλά και άλλων δύο αδελφών οργανώσεων. Ε, ο στόχος μας ήταν να διασφαλίζουμε τη συνεργασία για διάφορα θέματα που αφορούν τις ε, ακτές. Αυτή τη στιγμή ένα κομμάτι του προπολογισμού μας αφορά τη συνεργασία με τις ε, λιμενικές ε, υπηρεσίες. Αν μας ενδιαφέρει να διασφαλίσουμε τη συνεργασία, πρώτα απ' όλα εμείς ε, είμαστε το κέντρο των πληροφοριών στον θαλάσσιο τομέα. Τις πληροφορίες που έχουμε τις ανταλλάσσουμε ε, βεβαίως μέσω ηλεκτρονικού τρόπου κυρίως. Δίδουμε τις πληροφορίες ε, στη Frontex ε, που και αυτή τις χρησιμοποιεί για δικούς της λόγους. Το ίδιο ισχύει και με την ΕΦΚΑ. Παίρνουμε πληροφορίες βέβαια και από αυτούς τους δύο εταίρους. Πέρα από αυτό, επειδή εμείς είμαστε πρωτοπόροι, χρησιμοποιούμε τα drones για διάφορους λόγους. χρησιμοποιούμε τα drone και για παρακολούθηση στη Μεσόγειο. Η Frontex χρησιμοποιεί τα drones για να κάνει και αυτή να επιτελεί το καθήκον της. Άρα, είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα συνεργασίας. Κατά τα άλλα, η ΕΦΚΑ στο χαρτοφυλάκιό της έχει τα σκάφη για ε, ναυτιλιακές επιθεωρήσεις και έχουμε εξοπλίσει ε, τα δικά τους σκάφη με μικρά drones τα οποία τους βοηθούν να ε, επιτελούν, όπως σας είπα, τους, το καθήκον τους να κάνουν τους ελέγχους, αλλά πέρα από αυτό, ε, εφόσον ε, εντοπίσουν πετρελοκυλίδες ή κάτι που εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας, μπορούν και εκεί να δραστηριοποιηθούν και έτσι και εμείς διαφυλάσσουμε τα χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογούμενου. Υπήρξε και μία ερώτηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ναυτιλία, την χρήση σκαφών, ε, την χρήση ε, σημαίων, ε, σημαίες ευκαιρίας τις αποκαλούμε. Παλαιότερα, πολλοί χρησιμοποιούσαν σημαίες ευκαιρίας Λιβερίας, Παναμά, τρίτων κρατών δηλαδή. Αυτή η τάση όμως έχει αλλάξει για πάρα πολλούς λόγους. Ένας εξ είναι ότι στην Ευρώπη Πλέον ναι, υπάρχει κάποια ευαισθητοποίηση για θέματα φορολογίας ε, και έτσι ε, τα σκάφη επανέρχονται στην Ευρώπη. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού πλέον στην Ευρώπη έχουμε ένα καλύτερο δίκτυο και έχουμε και ένα καλύτερο ρόλο ε, του ΕΜΣΑ στον έλεγχο των λιμανιών. Έχουμε το πρόγραμμα ΘΕΤΙΣ, το οποίο επιτρέπει να εντοπιστούν τα ίδια εργαλεία, τα ίδια κριτήρια ε, για τον εντοπισμό των σκαφών και για την ανταλλαγή πληροφοριών στα σκάφη που ελέγχονται σε ευρωπαϊκά λιμάνια. Άρα δηλαδή έχουμε τις ίδιες συνθήκες εργασίας, ε, για τα σκάφη τα οποία λιμενίζονται σε ευρωπαϊκά λιμάνια. Προηγουμένως ε, ετέθη ένα ερώτημα για την ε, ναυτοσύνη γενικότερα. Ο δικός μας ο ρόλος είναι να στηρίζουμε τα κράτη-μέλη στην ε, εφαρμογή παγκόσμιων προτύπων στα ευρωπαϊκά ε, σκάφη αλλά και στα ευρωπαϊκά λιμάνια και είμαστε περήφανοι που στις αρχές του επόμενου έτους στον ΕΜΣΑ θα φιλοξενήσουμε ένα workshop ε, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε να προάγουμε την εφαρμογή ε, αυτού του τόσο σημαντικού εργαλείου για την Ευρωπαϊκή Ναυτιλία αλλά και γενικότερα για τον κόσμο. Θα μπορούσα να συνεχίσω, αλλά δεν ξέρω αν απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Κύριε Ρικέ, θέλετε να απαντηθεί η ερώτησή σας. Απαντήστε παρακαλώ στην ερώτηση του κύριου Ρικέ, αν δεν με πατάει η μνήμη μου. Θέλω να ξέρω τι μας... Ποια είναι υπερπεριφερειακές, τις υπερπεριφερειακές περιοχές, τις υπερπόντιες περιοχές. Ναι, ήταν το ερώτημα τις υπερπόντιες περιοχές που είχα θέσει. Well, in that context I said, um, if and when requested by the member... Όταν και αν το ζητήσουν τα κράτη-μέλη. Εμείς ε, αναπτύσσουμε τις δυνάμεις μας, παρακολούθηση μέσω του δορυφόρου, χρήση. Ε, η χρήση του δορυφόρου μας επιτρέπει να εντοπίσουμε και να ελέγχουμε την κυκλοφορία παγκοσμίω. Ε, οπουδήποτε λοιπόν και οποτεδήποτε μας το ζητήσουν τα κράτη-μέλη, εμείς αναπτύσσουμε τα μέσα μας. Από εκεί και πέρα διαχειριζόμαστε μια σειρά από project Διεθνού χαρακτήρα, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα. Εντάξει, δεν έχει σχέση με αυτό που είπατε ε, με τα υπερπόλια μερίσματα δηλαδή, αλλά έτσι εξασφαλίζουμε εμείς ε, ένα ίσο πεδίο ευκαιριών. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ για όλες τις απαντήσεις. Να ευχαριστήσω την κυρία Μάρκοβιτς Κόστελατς. Ε, είναι ένα ζήτημα το οποίο μόλις αρχίζει, έτσι, μόλις ανοίγει, θα υπάρξει ένας οδικός χάρτης για τις θαλάσσιες μεταφορές οπωσδήποτε κατά τη διάρκεια αυτή της θητείας, ελπίζω έχουμε ήδη πολλές σχετικές εκθέσεις και βέβαια θα επικεντρωθούμε στη συνέχεια ε, και στην κλιματική πρόκληση και στην ψηφιακή πρόκληση με συγκεκριμένους στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν διότι ο χρόνος είναι μετρημένος και πρέπει και ο τομέας θαλάσσιων μεταφορών ε, να πάρει θέση και να προσαρμοστεί και αυτός με βάση τον οδικό χάρτη. Ε, και αυτό αφορά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Θα πρέπει με δραστικό τρόπο και κάπως ριζικό ε, να, συνοδεύσουμε αυτή την προσπάθεια αν θέλουμε να σεβαστούμε τις συμφωνίες των Παρισίων. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Είστε πάντα καλοδεχούμενοι σε αυτή την Επιτροπή Μεταφορών. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να ξαναέρθουμε στη Λισαβόνα να σας συναντήσουμε διότι είναι πάντα καλό να ε, επισκέπτεται κανείς τις υπηρεσίες να πηγαίνει επί τόπου ε, προλέπετε άλλωστε στην ημερήσια διάταξη για το 2020 να σας επισκεφτούμε λοιπόν διακόπτουμε για 6 λεπτά 6 λεπτά στη συνέχεια έχω μια σειρά από οικονομικά ζητήματα. Θα δούμε μια μελέτη ε, πραγματικά συναρπαστική. Θα μας μιλήσει για το σύνολο των επενδύσεων που θα έπρεπε να είχαν γίνει ή που, θα, ή που πρέπει να γίνουν και το σύνολο των δημοσιονομικών ε, φακέλων σε έξι λεπτά. Έχετε χρόνο για ένα καφέ νομίζω. Τα λέμε.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 Mes chers collègues, nous allons reprendre notre, nos travaux, s'il vous plaît. Συνάδελφοι, ξαναρχίζουμε τις εργασίες μας. Παρακαλώ, πάρτε θέσεις. Λοιπόν, θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της μέσης διάταξης. Θα εξετάσουμε τη μελέτη του, του θεματικού τμήματος για τη χρηματοδότηση των project. Κύριε Βιμ Βαντενκάμπ, δεν αλλάζει ο κ. Βαντενκάμπ. απαράλλαχτος. Λοιπόν, θα περάσουμε στη μελέτη του θεματικού τμήματος για τα project στον τομέα των μεταφορών. Θέλουμε εδώ να αναδείξουμε τα διάφορα οικονομικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα για αυτά τα project. FEDER, Μηχανισμός Διασύνδεσης, Εύση οι μεταφορές ε, και η σχετική πολιτική η ευρωπαϊκή εξαρτάται από αυτά. Χαίρομαι που έχουμε εδώ δύο εμπειρογνώμονες μαζί μας, τον Χωσέ Μανουέλ Βασαγιό, ο οποίος είναι καθηγητής στο τομέα των μεταφορών στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο της Μαδρίτης, και η Λάουρα Γκαρίδο, η οποία επίσης είναι καθηγήτρια ερευνήτρια στο Πολυτεχνείο της Μαδρίτης, είναι οι συντάκτες αυτής της μελέτης που θα μας παρουσιάσουν για 10 λεπτά Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η συζήτηση με τους βουλευτές μας. Έχετε τον λόγο. Θέλω να είμαι σαφής τώρα εδώ για το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας ε, για να μείνει και χρόνος ε, για συζήτηση μετά. Hear me? Ευχαριστώ. Με ακούτε? Very much, ladies and gentlemen, members of... Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ που μου δίδετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τη μελέτη την οποία κάναμε. Μας την ανέθεσε η Πετροπή Τραν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Λάουρα Γαρίδο που κάθεται δίπλα μου. Φτιάξαμε αυτή τη μελέτη και θα απαντήσει και σε κάποιες απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα, για να δούμε κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν. Ποια είναι η παρούσα κατάσταση της χρηματοδότησης. Είναι αποδοτική, είναι κατάλληλη. Δεύτερον, για να δούμε πώς διαγράφεται το μέλλον. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ανοιχνεύσουμε ειδικές, ε, ειδικούς τομείς ενδιαφέροντος για το των μεταφορών, να αναλύσουμε τις μελλοντικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή και να παρουσιάσουμε νέες ιδέες ε, βελτίωση οργανωτική και συστάσεις στα πλαίσια του νέου πολυετούς χρηματοδητού. Πρώτα απ' όλα, ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι, τρεις είναι οι κύριοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την πολιτική στον τομέα των μεταφορών. Πρώτα απ' όλα, να δημιουργήσουμε συνεκτικότητα. Δεύτερον, να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και να συμπληρώσουμε το ten Εδώ έχετε την ε, χάρτη της Ευρώπης. Τρίτον, να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις σε θέματα στρατηγικής κινητικότητας. Ψηπιοποίηση, ε, εγκατάλειψη του άνθρακα, ασφάλεια, ε, κινητικότητα στον τομέα των στο στρατιωτικό κλάδο. Πρώτα απ' όλα, ας ταξινομήσουμε τα μέσα τα οποία διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πρώτα απ' όλα την, ε, χρηματοδο... την ε, επιχορηγήσεις, τα δάνεια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και νέα καινοτόμα χρηματοπιστωτικά μέσα. Δεύτερον, ποια είναι τα σχέδια, τα project που υποστηρίζονται τα TNT ή και κάποια άλλα project, ποια είναι η προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση, η διαχείριση από κοινού. Αυτό αφορά τα Ταμείο Συνοχής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, σημαίνει ότι συμμετέχουν στα διαχείριση τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη έχουν πάρα πολύ μεγάλη ελευθερία τη διαχείριση των τελειών. Δεύτερον, έχουμε άμεση χρησιμοποιητοποίηση, ε, ε χρημα, ε, διαχείριση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΙΝΕΑ. Ε, και τρίτον, έχουμε άλλα, B και άλλα. Ποιες είναι οι προτεραιότητες πολιτικής. Έχουμε το Ταμείο Συνοχής, το ΦΕΝΤΕΡ που είναι ταμεία κυρίως για την συνοχή και η διαχείρισή τους γίνεται από κοινού. Διαχειρίζονται ε, τα τεντά ε, και άλλες δυνατότητες σε περιφερειακό επίπεδο. Επίσης έχουμε το ΣΕΦ, Connecting Europe Facility, το μηχανισμό συνδέοντα στην Ευρώπη και έχουμε ανάλογα βλέπετε όπως βλέπετε σε αυτό τον πίνακα πώς γίνεται η διαχείριση των μέσων των χρηματοδοτικών. Όλα εξαρτώνται σε αυτή την περίπτωση και από την ε, προστιθέμενη αξία, από την ε, δυνατότητες της κινητικότητες και τι είδους ε, Κονδύλια έχουμε εδώ πέρα, επιχορηγήσεις, δάνεια και κυρίως εδώ πέρα είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επιδείξεων που τα χειρίζεται. Θα ήθελα τώρα να μιλήσω για τις τάσεις που διαγράφονται. Τα παραδοσιακά μέσα όπως το Ταμείο Συνοχής βλέπουν να μειώνονται τα κονδύλια τους. μέσα όπως το ΙΣΕΦ, δηλαδή το ΣΕΦ, το Μηχανισμό Συνδέοντας την Ευρώπη για τις μεταφορές, δεν βλέπει να φτάνουν τα κονδύλια του σε σχέση με τα προηγούμενα χρηματοδοτικά πλαίσια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλο και περισσότερο ενθαρρύνει τη χρησιμοποίηση καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων παρά επιχορηγήσεων. Ας συνεχίσουμε εξετάζοντας ποια είναι τα θέματα και ποιες είναι, ποια είναι τα επιτέγματα όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων. Θα κάνουμε κάποιες ερωτήσεις και η πρώτη είναι όλα αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν οριστεί σωστά σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα, σύμφωνα με την ε, ΕΚΑ πρέπει να στοχοποιηθούν περισσότερο. Και το Ταμείο Συνοχής και το ΦΕΝΤΕΡ πολλές φορές δίδουν τα κονδύλια στα κράτη-μέλη, τα οποία τα δίδουν με τη σειρά τους σε προτεραιότητες ε, περιφερειακού επίπεδου. Στο θέμα των αεροδρομίων, των περιφερειακών που μελετήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να χρησιμοποιεί το μείωση για να βελτιωθούν τα μικρά αεροδρόμια, τα περιφερειακά, σε μικρές ε, πόλεις, μεταξύ άλλων. Ποια είναι τα θέματα που υπάρχουν και ποιες είναι οι επιτεύξεις. Τα ποσά που δίδονται καλύπτουν τις όλο και αυξανόμενες ανάγκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβλέπετε ότι δεν είναι αρκετά τα κονδύλια τα οποία γίνονται στο ΣΕΦ. Βλέπετε πώς εξελίσσονται τα προγράμματα σε δις από το 2014 μέχρι το 2020 βλέπετε ότι υπήρξαν στα τελευταίο χρηματοδοτικό πλαίσιο ε, αρκετά κονδύλια, αλλά υπήρχαν και σχέδια που δεν καλύφθη. Το επόμενο θέμα. Ε, ο, είναι ισοσκελισμένη η κατανομή αυτών των κονδυλίων ε, ανάλογα με τις περιοχές. Πολλές φορές κάποιες καινοτόμες προσεγγίσεις είναι πάρα πολύ ε, πολύπλοκες για κάποιες αναπτυσσόμενες περιοχές. Πρόκειται για καλά μέσα, αλλά οποία δύσκολα μας μπορούν να, να εφαρμοστούν σε περιοχές που δεν έχουν την κατάλληλη ανάπτυξη. Δεύτερον, είναι κατάλληλη η διαδικασία αξιολόγησης. Ε, μία από τις κυρίες επικρίσεις είναι ότι δεν υπάρχει εστιασμός στα αποτελέσματα και στον αντίκτυπο. Και πρέπει να γίνει η κατάλληλη αξιολόγηση ακόμη και από το ε, ελληνικό συνέδριο. Τρίτη ερώτηση είναι αποτελεσματικά συντονισμένα όλα αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ακόμη κάποιες επικαλύψεις και υπάρχουν κάποια παραδείγματα περιορισμένης δράσης. Όλες οι διοικητικές ε, διαδικασίες πολλές φορές μπορούν να αποτελέσουν ε, εμπόδιο. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Στη... Μπορούν τα διοικητικά θέματα να βελτιωθούν. Μελετήσαμε μία διασυνοριακή HSR σύνδεση. Είδαμε ότι είχε επιλεχθεί το project αυτό ε, για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ποσοστό 40%. Υπήρχε όμως από μία από τις αφορόμενες περιοχές μεγάλη αντίθεση, άρα δεν μπόρεσαν να γίνουν ε, οι κατάλληλες ε, επενδύσεις και να μπορέσει να μελετηθούν σωστά οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις για να αναπτυχθεί αυτό το project παρά το γεγονός ότι είχε ε, επιλεγή. Υπάρχουν δυνατότητες και υπάρχουν προκλήσεις για το μέλλον και πρέπει να τις εντοπίσουμε ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την όλη κατάσταση. Βασικά εντοπίσαμε ότι υπάρχουν ακόμη αρκετά θέματα τα οποία δεν έχουν επιληθεί. Το θέμα της πολυτροπικότητας θα μπορούσα να σας πω ότι έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα, αλλά δεν το λύσαμε ακόμη. Επίσης, να υπάρχει το ίδιο επίπεδο μεταχείρισης, επίπεδο φορολογία κτλ. Και το θέμα της ασφάλειας επίσης είναι σημαντικό. Υπάρχουν επίσης άλλε αναδιόμενες ε, ε, δυσκολίες και προκλήσεις, η κλιματική αλλαγή, η μόλυνση, η βιοπικιλότητα, η ανθεκτικότητα, τάσεις που διαγράφονται στις διάφορες περιοχές όσον αφορά την, ε, τους κατοίκους, δηλαδή έχουμε αύξηση της ε, αστι... Ε, αστικές περιοχές, έχουμε διάφορες περιοχές οι οποίες είναι απομονωμένες, από τις οποίες φεύγει ο κόσμος και έχουμε γυράσκοντα πληθυσμό. Επίσης υπάρχουν, υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε. Ποιες είναι οι συστάσεις μας για τη χρηματοδότηση. Θα πρέπει να αυξηθούν τα κονδύλια τα οποία δίδονται για τις ανάγκες των μεταφορών, κυρίως στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχής και του Μηχανισμού Συνδέας στην Ευρώπη. Επίσης, να αυξηθούν τα κονδύλια τα οποία δίδονται για την προσαρμογή της, ε, ε, των υποδομών για να καλυφθούν νέες ανάγκες κινητικότητας. Να δοθεί προτεραιότητα σε μέτρα που προγάγουν την ε, ε, διαλειτουργικότητα και την ενσωμάτωση και να μπορέσει να ιεραρχήσουμε τις ε, προτεραιότητες στις μητροπολιτικές περιοχές και στις περιοχές που έχουν προβλήματα ανάπτυξης. Δεύτερο, δεύτερο τμήμα συστάσεων για την οργάνωση. Για να δοθεί χρηματοδότηση στα κράτη-μέλη θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε διασυνοριακά τμήματα και περιοχές. Εάν λοιπόν δεν κάνετε κάτι το οποίο είναι ε, κοινού ενδιαφέροντος, δεν θα χρηματοδοτήσετε πλέον. Δεύτερον, να συνδυάσουμε περισσότερες ευέλικτες προσεγγίσεις για το συνδυασμό ε, οικονομικών πόρων. Τρίτον, να φτιάξουμε ένα κοινό πλαίσιο αξιολόγησης για όλα τα project στον τομέα των μεταφορών που υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δώσουμε σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για ε, καινοτόμα μέσα στα πλαίσια του InvestEU. Και να ομοιογενοποιήσουμε και να απλοποιήσουμε τις διοικητικές διαδικασίες. Το θέμα τώρα της διαχείρισης. Θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε μία ε, αξιολόγηση του κοινού πλαισίου ανεξάρτητη για όλα τα project τα οποία χρηματούν την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουμε μία ενιαία, έναν ενιαίο ευρωπαϊκό οργανισμό μεταφορών. Να παρέχουμε τις, κατάλληλες τις κατάλληλες, ε, την κατάλληλη μελέτη και συμβουλή σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και να μπορέσουμε να προωθήσουμε την εναρμόνιση των τελών της φορολόγησης και των επιχορηγήσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ε, παρουσίασή σας. Υπάρχουν πολλά θέματα του προπολογισμού που τα γνωρίζουμε, όπως ξέρετε. Έτσι, κύριε Ρικέ. Λοιπόν, να ξεκινήσει τώρα η συζήτηση. Κύριε Μαρινέσκου, Είστε και εσείς από τους εμπειρογνώμονες ε, του Μηχανισμού Διασύνδεσης, είστε από τους εισηγητές μας, έχετε το, δίκ, το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση, αυτή την έκθεση. Μου άρεσε αυτή η πρώτη σύσταση να αυξηθεί η χρηματοδότηση. Αν μπορείτε να μιλήσετε με το Συμβούλιο, ε, πείτε τους ε, ε, δείτε τι έχουν κάνει αυτοί εκεί στη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση με τα κονδύλια αυτά. Εδώ και καιρό ασχολούμαι με την πραγματική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των Ευρωπαϊκών Ταμείων σε σχέση με τις μεταφορές. Θέλω δηλαδή να δω ένα χάρτη με τους διάφορους διαδρόμους των Ευρωπαϊκών Δικτύων, τα project που έχουν χρηματοδοτήσει ε, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, ο, από όλα τα ταμεία, ταμείο συνοχής, ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης, πού πήγαν τα χρήματα πού επενδύθηκαν και ποιο είναι το ποσοστό αποτελεσματικότητας. Και αυτό δεν το βλέπω εδώ. Αυτό θα βοηθούσε ιδιαίτερα από ό,τι κατάλαβα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επανεξετάσει ε, τον κανονισμό TNT θα βοηθούσε λοιπόν να ξέρουμε πώς επενδύθηκαν τα χρήματα αυτά. Κατά τα λοιπά, οι συστάσεις είναι καλές. Ε, δεν ξέρω πώς θα καταφέρετε να έχετε μία και μόνο υπηρεσία. Ωραία θα ήταν. Αλλά να βάλετε μαζί τώρα το σιδηρόδρομο ε, και την ε, αεροπορία για την αεροπορία δεν υπάρχει, έτσι, υπάρχει η ΆΣΑ. Η ΆΣΑ ασχολείται με την ασφάλεια όμως μόνο. Και πρόκειται για σύμπραξη. Θέλετε να πάρει το σιδηρόδρομο μαζί με τις θαλάσσιες ε, μεταφορές. Ε, τους ρωτήσατε, ρώτησατε αυτές τις υπηρεσίες να ακούσετε και μία άποψη. Ίσως και την ΙΝΕΑ. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολο. Η συντήρηση των υποδομών. Αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο συναντούμε συχνά τα τελευταία, τελευταία χρόνια. Είναι αλήθεια ότι θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί αυτό από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Θα ήταν όμως και κάπως υπερβολικό. Έτσι, πριν από 10 χρόνια περίπου χρηματοδοτήσαμε τη δημιουργία νέων υποδομών, τώρα για τη συντήρησή τους, ε, εντάξει, κάπως υπερβολικό μου φαίνεται. Χρειαζόμαστε χρήματα για νέα στοιχεία που θα συμπληρώσουν αυτούς τους διαδρόμους. Ε, αυτός πρέπει να είναι ο βασικός αποδέκτης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Από εκεί πέρα τα κράτη-μέλη μπορούν να εργαστούν γύρω από το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Μαρινέσκου. Η κυρία Γκαρσία Μουνιώθ έχει το λόγο. Ναι, από την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση που ήταν και πλήρης. Εγώ υπερασπίζομαι την έξι, τις έξυπνες μεταφορές που σέβονται το περιβάλλον. Είναι καλό λοιπόν να επενδύσουμε στο σιδηρόδρομο αλλά και στους λιμένες έτσι ώστε η μεταφορά και επιβατών αλλά και πορευμάτων να γίνεται κατά προτεραιότητα είτε με τρένο είτε με πλοίο. Βεβαίω δεν μπορούν να γίνουν όλα, όλες οι μεταφορές με αυτά τα μέσα. Θα αυξηθεί κατά 80% το εμπόριο, το, το, το, το, η μεταφορά εμπορευμάτων και ένα 40% των επιβατών. Οπότε ε, εξακολουθεί ο τομέας ε, αυτός των θαλάσσιων μεταφορών ε, να είναι ο να έχει την πρωτοκαθεδρία. Θα πρέπει να προσέχουμε βεβαίω που επενδύουμε, να είμαστε αποτελεσματικοί. Είμαστε ταυτόχρονα ανοιχτοί και σε νέε καινοτόμε λύσει. Και εδώ έρχεται το ερώτημά μου. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν αναλύσει ε, για το τι είδου επενδύσει σε υποδομέ οδηγούν σε μεγαλύτερα ωφέλη για την κοινωνία με βάση την υπάρχουσα, τον υπάρχον τρόπο ζωή, αν θέλετε. Λαμβάνοντα όμω ταυτόχρονα υπόψη και του κλιματικού στόχου που έχουμε θέσει για του οποίου έχουμε δεσμευτεί. Πρέπει να προσαρμοστούμε στι ανάγκε κινητικότητα στο μέλλον. Η κινητικότητα έχει να κάνει με τι αναλυτικέ ε, πηγέ καυσίμων, ε, το πρασίνισμα. Ε, αυτά επηρεάζουν ιδιαίτερα τις μεταφορές τις οδικές. Ο κύριος Μπαθαντία θα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το πρώτο που θα ήθελα να πω εγώ ε, είναι να συγχαρώ αυτή την ομάδα που συνέταξε αυτή την έκθεση. Είναι πολύ σαφής ε, και συγκεκριμένο, συγκεκριμένη έκθεση αυτή. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα θέμα, το θέμα της ε, στρατιωτικής κινητικότητας. Το 2017 η Ισπανία έστειλε περίπου 551 στρατιώτες, 15 οχήματα, ε, Καναντέρ ε, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους γείτονές μας, ε, τους Πορτογάλους, το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές τους. Αυτό είναι ένα παράδειγμα στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ δύο κρατών μελών όπου κατέστη σαφές εδώ και ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική αποτελεσματικό το έργο των δυνάμεών μας βοηθώντας τους Πορτογάλους φίλους. Γιατί το λέω αυτό, διότι όταν μιλάμε για στρατιωτική συνεργασία για να αντιμετωπιστούν φυσικέ καταστροφές και συστήματα πολιτικής άμυνας, πρέπει να μιλήσουμε και για την μεταφορά. Διότι οι μεταφορές είναι σημαντικές για την αποτελεσματικότητα ε, όλων αυτών των επεμβάσεων σε, όλα, σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Υπάρχει όμως ένα βασικό εμπόδιο στις μεταφορές αυτές είναι η έλλειψη υποδομών στον τομέα των μεταφορών για να, μεταφερθούν τέτοιου, να μεταφερθεί τέτοιο εξοπλισμό μεταξύ κρατών μελών. Ε, έτσι λοιπόν αυτή η έκθεση είναι πολύ ε, χρήσιμη. Θέλω να ευχαριστήσω ε, που ανταποκριθήκατε στο αίτημα αυτής της Επιτροπής και να πω ότι για πρώτη φορά, όπως είπατε κι εσείς, ο μηχανισμός Connecting Europe ε, προέβλεψε ε, ένα κονδύλιο για την επόμενη περίοδος ένα σημαντικό κονδύλιο για τα project αυτά που έχουν να κάνουν με την κινητικότητα στρατιωτικού υλικού για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού, ε, την, την στρατιωτική κινητικότητα δηλαδή. Και αυτό βεβαίως ε, συνάδει και με την ψηφοφορία ε, των μηχανισμών, την ψήφιση των μηχανισμών για το Connecting Europe. Αυτά τα σχέδια χρηματοδότηση είναι απαραίτητα όταν μιλάμε για τη συνεργασία στον τομέα τη άμυνα, για να είναι πιο γρήγορη αυτή η συνεργασία, να μην υπάρχουν εμπόδια και για να διευκολύνουμε τι δυνατότητε απάντηση απέναντι σε επίγουσε καταστάσει, φυσικέ καταστροφέ και βεβαίω όταν υπάρχουν ανθρωπιστικέ κρίσει. Περισσότερο από ποτέ λοιπόν είναι σημαντικό να προχωρήσουμε σε πολιτικές άμυνας, κοινέ πολιτικές άμυνας είναι απαραίτητο να επενδύσουμε ε, σε ε, τρόπους μεταφοράς που διευκολύνουν τις στρατιωτικές μεταφορές στην Ευρώπη. Ε, χαίρομαι λοιπόν που μέσω αυτής της Επιτροπής μπορέσαμε να πετύχουμε η έκθεση αυτή να τεθεί επιτάπητος και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα συνεισφέρει για να βελτιωθούν οι σχέσεις αλλά και οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Για άλλη μια φορά συγχαρητήρια σε εσά. Ευχαριστώ κύριε Μπάουθα Ντίαθ. Ε, μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με αυτό που είπατε θα θέλω να αναφέρω. Το σχέδιο κινητικό, το Ταμείο Κινητικότητα, μιλάμε για military mobility, έτσι, στρατιωτική κινητικότητα. Και λέτε, όλα τα οποία αναφερθήκατε, ε, με τι πυρκαγιέ, είναι ανθρωπιστικέ, έτσι, ανθρωπιστικού περιεχομένου. Γι' αυτό λοιπόν θα ήταν καλύτερο να μιλήσουμε για Ταμείο στρατιωτικής και ανθρωπιστικής κινητικότητας. Αυτό το και ανθρωπιστικής δεν πέρασε. Ενώ το Ταμείο θα έχει αυτή τη χρειά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας και θα πρέπει να το επιλύσουμε τους επόμενους μήνες. Ε, κύριε Κυριάνκοφ, έχετε το λόγο. Ε, κύριος μάλλον. Ναι, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο ε, συντάκτες της έκθεσης, ε, την κυρία Γκαρίδο και τον κύριο Βασαγιό. Πραγματικά είμαι εντυπωσιασμένο. Είναι πολύ συγκεκριμένο, ε, πολύ ακριβές, ε, ταυτόχρονα λαμβάνει μια πολύ σημαντική συνάντηση με σήμερα, συνάντηση με τη δική μας, πολύ πιο σημαντική, στη Μαδρίτη, COP25 και συνδέεται με την παγκόσμια πρόκληση που έχουμε να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων που προκλούν το δεξιό του άνθρακα. Ε, εσείς λέτε ότι χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για τις μεταφορές. Είστε και δύο μηχανικοί από όσο ξέρω, έτσι. Ως μηχανικοί, φαντάζομαι ότι συναντήσατε συχνά το θέμα της ζήτησης που προκαλείται. Όταν δηλαδή κατασκευάζουμε κάτι, θα μας τα ζητηθεί θα χρησιμοποιηθούν περισσότερο υποδομέ. Δεν ανησυχείτε λίγο ότι αυτή η κούρσα προ περισσότερε υποδομέ θα οδηγήσει σε περισσότερε μεταφορέ και σε περισσότερε εκπομπέ τελικά. Βεβαίω ε, να μιλήσουμε για τα τεχνικές λύσεις, ε, για την, την ηλεκτρική ενέργεια, την τρίτη γενιά βιοκαυσίμων, ε, τη διαχείριση της ζήτησης. Όμως τελικά δεν θα πρέπει να το δούμε και ευρύτερα το θέμα του ευρύτερου δηλαδή περιβαλλοντικού κόστους της μεταφοράς. Εάν έχετε κάτι να πείτε από αυτού θα, θα με ενδιαφέρε. Επίσης είναι κάπως ηρωνικό ότι η μόνη πραγματικά νέα μορφή χρηματοδότηση είναι η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, έτσι. Εντάξει, όπως είπατε και εσείς πρόεδρε, αυτές οι στρατιωτικές δαπάνες χρησιμοποιούνται έτσι ώστε στρατιωτικό προσωπικό να αντιμετωπίσει ακραία καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιές που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Μήπως λοιπόν θα ήταν καλύτερα απλά, απλά να έχουμε ένα, ένα ταμείο για το κλίμα που να, για να καλύπτει όλε αυτέ τι τεράστιε προκλήσει, είτε μιλάμε για πλημμύρε, είτε μιλάμε για πυρκαγιέ που έχουν σχέση με την κλιματική αλλαγή. Και υπάρχει ένα θέμα τελικά του πόσο ανθεκτικό είναι το δίκτυο μεταφορών σε αυτό το κλίμα και σε αυτό τον καιρό που θα βρούμε μπροστά μας όχι σε 25-30 χρόνια σε 5 χρόνια αλλά και με βάση κάποια καλοκαίρια και κάποιους χειμώνες που έχουν περάσει το τελευταίο δια, που, ζήσαμε το τελευταίο διάστημα όπου πραγματικά τα κρέα καιρικά φαινόμενα, καιρικά φαινόμενα οπωσδήποτε ε, σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Δέχεστε λοιπόν ότι υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ αυτών των περισσότερων υποδομών και, της, και των κλιματικών στόχων. Έχετε κάποια σκέψη για το πώς μπορούμε αυτό το κόστος ε, να το συνυπολογίσουμε. Σκεφτείτε τις, τις προτεραιότητες σε επίπεδο χρηματοδότησης. Δαπανίστε τουλάχιστον σε βιώσιμες μορφές μεταφορών. Όχι απλά να διαβρύνουμε δίκτυα για να έχουμε όλο και περισσότερες μεταφορές ε, με χρήση άνθρακα. Ευχαριστώ κύριε Κόφο. Κύριος Ζήλε έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την παρουσίαση της έκθεσης. Ε, πολύ καλή. Ε, η παρουσίαση τουλάχιστον, δεν έχω διαβάσει το έκθεση. Την έκθεση θέλω να κάνω πρώτα κάτι, κάποια ερωτήματα σαν και αυτά που ανέφερε ο κύριος Μαρινέσκου. Έχουμε το Connecting Europe Facility, το σχετικό Ταμείο είναι σχεδόν 15 χρόνια. Έτσι, δύο συνεχόμενες θητείες. Μήπως πρέπει η Κομισιόν ε, είναι, η χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή σχετίζεται με το Connecting Europe και ζητούν οι φορολογούμενοι, ρωτούν τελικά ολοκληρώθηκαν τα project αυτά. Ποια ολοκληρώθηκαν κάποια ε, βεβαίως project έχουν προθεσμία 2026, αλλά ε, αργότερα κάποιες εμβληματικές πρωτοβουλίες, κάποια εμβληματικά project. Ιδιαίτερα για τις χώρες του Ταμείου Συνοχής, ε, ε μήπως θα πρέπει η Κομισιόν να προετοιμάσει την ανάπτυξη του κάθε ε, διαδρόμου, πόσα χρήματα έχουν δαπανηθεί για του κάθε διάδρομο. Κάποια κράτη-μέλη έχουν διασυνοριακά project, ε, χρησιμοποιούν χρήματα από το Ταμείο Συνοχή, αλλά αυτό δεν ταιριάζει με τι απαιτήσει ε, για το Connecting Europe ε, που έχουν να κάνουν με την ταχύτητα του δρόμο κτλ. Οπότε ουσιαστικά χρήματα χάνονται και κάποια χρήματα ε, των, του Ευρωπαίου Φορολογούμενου. Μπορούμε πρέπει να ρωτήσουμε, να ζητήσουμε από την Κομισιόν με βάση την έρευνά σα να το εξετάσει αυτό. Επίση υπάρχει και μια σύγχυση με αυτό που μόλι άκουσα, ότι ενδεχομένω θα χρειαζόμαστε λιγότερε υποδομέ. Τι θα πει αυτό. Η Ευρώπη είναι μεγάλη, έτσι. Είναι, ποικίλουν οι καταστάσει. Μεταξύ χωρών τη Βαλτική ε, και του κέντρου τη Ευρώπη δεν υπάρχει καμία διασύνδεση με σιδηρόδρομο. Καμία. Και ο σιδηρόδρομο ε, ε, βεβαίω παράγει πολύ λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα. Είμαστε λοιπόν πολύ ευάλωτοι σε κάποιους τομείς. Να πούμε, αν πούμε δηλαδή θα σταματήσουμε να φτιάχνουμε υποδομές, ιδιαίτερα για τα project που έχουν να με τους διαδρόμους, θα ήταν τελείω λαθασμένο αυτό. Υπάρχει ένα θέμα κινητικότητας, έτσι. Δεν, υπάρχει, δεν υπάρχει μόνο θέμα περιβάλλοντος. Υπάρχει ε, και μια γειτονία στα ανατολικά, όπου υπάρχουν χώρες οι οποίες ε, ε εισβάλλουν ε, σε άλλες χώρες. Λοιπόν, direct management τώρα, άμεση ε, διαχείριση. Πόσο μακριά πρέπει να πάμε, διότι για το Connecting Europe Facility ε, ε, έχουμε κάποιες άμεσες, κάποια άμεση διαχείριση, αλλά υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του η νέα και των εθνικών αρχών στα διασυνοριακά project. Τι μπορεί να γίνει για να υπάρξει βελτίωση, θα χαθεί χρόνος. Θα, θα έχουμε διαδικασίες δημοσίων προμηθειών, ε, Άχρηστε, Θα δυσκολευτούμε να διαχειριστούμε αυτά τα project ε, όπου εμπλέκονται τρει και τέσσερι και πέντε χώρες. Έχετε ιδέες για το πώς μπορούμε να το εξορροπήσουμε αυτό, τι τις εξουσίες δηλαδή της η νέα ε, και τι εξουσίες των εθνικών αρχών εφαρμογής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζήλε. Η κυρία Κουντουρά έχει το λόγο, παρακαλώ. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντάκτες της έρευνας. Η αλήθεια είναι ότι διαβάζοντας ε, τη μελέτη σας απογοητεύτηκα καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ καταλήγεται ότι οι σημερινές πολιτικές δεν έχουν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικές ανισότητες. Και ενώ οι ανάγκες είναι τεράστιες, όπως πολύ σωστά επισημαίνεται, το Συμβούλιο θέλει να κόψει τους μελλοντικού πόρους για την πολιτική συνοχής Βρισκόμαστε όμως σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Από τη μία είναι η πρόκληση της κλιματικής κρίσης και από την άλλη το τόσο σημαντικό δημογραφικό ζήτημα το οποίο σπάνια ακούγεται εδώ στις Βρυξέλλες και ειλικρινά θέλω να σας ευχαριστήσω που το θίγετε έστω και επιγραμματικά σε συνάρτηση με τις πολιτικές μεταφορών. Η κλιματική πολιτική Έρχεται λοιπόν στο προσκήνιο και σχεδιάζουμε τις υποδομές μας τα τελευταία δέκα χρόνια σε ορίζοντα τριακονταετίας και πεντηκονταετίας και σε μεγάλο βαθμό με πολύ παλιά εργαλεία και ανεξάρτητα από τις κλιματικές πολιτικές που θα αλλάξουν δραματικά πολλές πτυχές της ζωής μας. Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω, θα είναι συμβατές οι υποδομές αυτές με τις κλιματικές μας δεσμεύσεις και τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις και αν όχι θα αναγκαστούμε σε 10-20 χρόνια να μειώσουμε απότομα τις μεταφορές επιβατών, εμπορευμάτων για να σώσουμε τον πλανήτη. Τα ερωτήματα αυτά είναι ζωτική σημασία, ίσως όχι τόσο για την κεντρική Ευρώπη, αλλά σίγουρα για τα περιφερειακά κράτη και ιδιαίτερα για τις απομακρυσμένες περιοχές που βλέπουν τον πληθυσμό τους να συρρυκνώνεται και κυρίως τα νησιά μας που αποτελούν μάλιστα κριτικές περιοχές με γεωστρατηγική σημασία Ήδη σήμερα οι νησιωτικές περιοχές, συχνά απομονωμένες, απορροφούν ένα δυσβάστακτο κόστος για τις μεταφορές από τους επιβάτες μέχρι τα βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα, νερό, ενέργεια. Η ζωή εκεί είναι δύσκολη, εκτός της θερινής περίοδου και αυτό φυσικά αντανακλάται στα δημογραφικά στοιχεία των περιοχών αυτών. Γι' αυτό το δεύτερο ερώτημά μου είναι εκτιμάτε ότι θα μπορούσαμε να θωρακίσουμε τις περιοχές αυτές και να εξασφαλίσουμε βιώσιμες και προσιτές μεταφορές με τα υπάρχοντα εργαλεία ή αν θα πρέπει να προσανατολιστούμε προς νέα και πιο στοχευμένα και πιο φιλόδοξα. Σας ευχαριστώ πολύ. Euh, ε, ευχαριστώ κυρία Κουντούρα. Ε, θέλουμε απαντήσεις στα ερωτήματά μας, οπότε οι ερωτήσεις οι επόμενες θα είναι σύντομες. Παρακαλώ, κυρία, ο κύριος Ρικέ, ναι, ευχαριστώ για αυτή τη μελέτη που είναι και ενδιαφέρουσα και πλήρης. Ε, τα συμπεράσματά της ε, πάνε άλλωστε προς την κατεύθυνση των ε, ε, ανησυχιών μας. Βεβαίως είναι συναγράφουμε στον Άγιο Βασίλειο. Ο Άγιος Βασίλης στην περίπτωση θεωρητικά είναι το Συμβούλιο, αλλά δεν είναι και τόσο γενναιόδωρος. Ε, το Συμβούλιο. Μιλάμε για σχέδια με ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία. Ε, θέλουμε να συμπληρώσουμε αυτό το δίκτυο, θέλουμε να βελτιώσουμε τις υποδομές των χωρών που αναπτύσσονται ακόμα και να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις, ψηφιοποίηση, ε, κλιματική αλλαγή, συντήρηση και αυτό με σημαντικούς δημοσιονομικούς περιορισμούς. Εσείς υπογραμμίζετε ότι η κεντρική διαχείριση τα χρήματα που διατίθενται, η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία είναι οι παράγοντες που επιτρέπουν να είμαστε αποτελεσματικοί σε δημοσιονομικό επίπεδο, ακόμα και αν οι πόροι είναι περιορισμένοι. Αυτό που εγώ διαπιστώνω είναι ότι τελικά πολλά από τα ταμεία αυτά την χάνουν αποκεντρωμένης διαχείρισης ή τη χάνουν διαχείριση από ενδιάμεσου, όπω η την χανουν διαχειριση απο ενδιαμεσου οπω η Επενδύσεων. Δεν πάμε προ επανασυγκέντρωση. αντιθέτω. Ε, πάμε προς αποκέντρωση. Και η πρόταση της ΕΦΣΗ είναι εξαιρετικά προβληματική, ε, διότι τελικά θα πάει σε χέρια που δεν είναι της Κομισιόν, ε, δεν πετύχαμε επανασυγκέντρωση εδώ ε, και έχει φανεί πολλές φορές ότι δεν λαμβάνει υπόψη την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων την Ευρωπαϊκή Προσταμένη Αξία στις επιλογές της, ιδιαίτερα στο κλιματικό επίπεδο. Πάμε δηλαδή προς μια επιδίνωση των μηχανισμών ελέγχου ε, και κατανομής, κάτι το οποίο ε, δεν συνάδει με αυτό που θέλετε εσείς. Επίσης δεν πάμε προς απλούστευση της ό,τι αφορά το διοικητικό σκέλος. Ε, δεν ξέρω αν είδατε τη σχέση του Συμβουλίου που ήταν καταστροφικό έτσι, για το Smart. τώρα το διαπραγματευτικό κουτί του Συμβουλίου είναι επίσης καταστροφικό αφού ακόμα και αυτό το κονδύλι για τα στρατιωτικά που πάλι θα κοπεί κατά 60% σχέση με το αρχικό ποσό, δεν ξέρουμε ποιο θα το διαχειρίζεται και πώ θα διαχειριστεί, διότι μιλάμε για τη δημοσιονομική γραμμή 5, την οποία δεν διαχειρίζεται αυτή η Επιτροπή. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν θα το διαχειρίζεται η Επιτροπή ή η νέα. Ε, οπότε, όπω καταλαβαίνετε, εδώ υπάρχει μεγάλη προχειρότητα. Σα ευχαριστώ πάντω για αυτή την έκθεση, η οποία περιλαμβάνει ακριβώ τι κατάλληλε συστάσει. Κάνουμε όμω το αντίθετο αυτή τη στιγμή και το μέλλον μου φαίνεται ζωφερό. Αυτό θέλω να πω σε μια εποχή όπου οι προκλήσεις ιδιαίτερα κλιματικέ είναι μεγαλύτερες από ποτέ. Λοιπόν, γράμμα στον Άγιο Βασίλη, αλλά ο Άγιος Βασίλης δεν είναι αυτός που νομίζουμε. Ε, σας ε, ευχαριστώ πολύ. Να πω και κάτι ακόμα. Ε, λυπάμαι που έχει μεταφραστεί αυτή η έκθεση μόνο σε μία γλώσσα της Ένωσης. Παρακαλώ όπως προβλέπουν οι θεσμοί μας, ε, να ζητηθεί να υπάρξει ε, μετάφραση σε τρεις γλώσσες της Ένωσης, τρεις γλώσσες εργασίας της Ένωσης, όπως προβλέπετε. Σας ευχαριστώ και για αυτή την τελευταία παρατήρηση. Θα το επαληθεύσω αν όντω η μελέτη αυτή πρέπει να γίνει σε, τρεις σε τρεις γλώσσες. Λοιπόν, από τον ε, καλό Άγιο Βασίλη ας περάσουμε στον κακό της παρέας. Δεν ξέρω αν πραγματικά έχουμε το δικαίωμα να είμαστε πιο αισιόδοξοι βλέποντας αυτή τη μελέτη που είναι εξαιρετική. Σας ευχαριστούμε και ως νέα Ευρωβουλευτής βλέπω ότι έχω πραγματικά εντοπίσει τα προβλήματα που έχουμε ως Πράσινη. ξέρετε ότι εμείς επιθυμούμε μεγάλες αλλαγές και στο τομέα των μεταφορών. Αν και δούμε τη μελέτη σας, βλέπουμε ότι αυτό είναι δύσκολο πραγματικά, διότι δεν ενεργούμε με το σωστό τρόπο. Περισσότερη εναρμόνεση και με το σωστό τρόπο. Είναι κρίμα το ότι μένουμε στις ιδέες του παλιού μας του κόσμου, αυτού που ξέραμε. Και μου αρέσουν και οι συστάσεις. Μιλάτε για μεγαλύτερη εναρμόνιση των επιχορηγήσεων, των τελών, της φορολόγησης. Όπως ξέρετε, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό το θέμα της ε, τιμολόγησης ή των ε, τελών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης υπάρχει το πρόβλημα της ε, αεροναυτιλίας, των μικρών αεροδρομίων. Καταλαβαίνετε ότι όλοι δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, δεν τη τις τη ίδια άρα είναι λανθασμένος ο τρόπο μα. Επίση, μιλάτε για ενιαίο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Μεταφορών. Δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη, αλλά κατά την άποψή μου, αυτό το οποίο ε, λείπει είναι να ασχολείται κάποιος με όλες τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον τομέα των μεταφορών. Ίσως ο καθένας θα πρέπει να ασχολείται με αυτά τα οποία πρέπει να κάνει. Δεν θέλουμε να αυξηθούν κατά πολλά ε, κονδύλια ο αλλά να αλλάξουν κάποια πράγματα. Είναι σωστά η δουλειά. Πιστεύω λοιπόν ότι εδώ στην ε, Επιτροπή μας θα κάνουμε την κατάλληλη πολιτική ώστε να αλλάξουν τα πράγματα και στην ε, μεταφορά, μεταφορά φρέτ και, και στο, για τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πολύ. για την μελέτη την οποία παρουσιάσατε και τα πορίσματά σας. Για τις διαφορές που υπάρχουν και γι' αυτό θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση σε σχέση με τις, ε, με τις ε, σιδηροδρομικές μεταφορές. Όταν κάνατε τη μελέτη σας, κάνατε σύγκριση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων περιοχών του κόλου. Υπάρχουν περιοχές άλλες που οι ιδιωτικές επενδύσεις ε, πηγαίνουν στην, στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Ξέρουμε ότι στο παρελθόν τα σιδηροδρομικά μας δίκτυα κάλυψαν πολλές υπήρους και τα 30 δις που έχουμε για την ε, συνδεσιμότητα καθώς και άλλα σχέδια που έχουμε δεν επαρκούν για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Χρειαζόμαστε 500 δις για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε με το σωστό τρόπο κάποιες περιοχές. Το ερώτημά μου λοιπόν το κύριο είναι μπορέσατε να κάνετε εσείς ε, μελέτη των συνδρομικές μεταφορές και ποια είναι η συνδρομή των ιδιωτικών επενδύσεων. Και μία άλλη παρατήρηση σε σχέση με τις προκλήσεις του άπειρων που μπορεί να είναι και ευκαιρίε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπατε ότι δεν έχουμε ούτε καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το κατάλληλο πλαίσιο που θα μας επιτρέπει να έχουμε δίκαιες συνθήκες ανταγωνιστικότητας μεταξύ των διαφόρων ε, τύπων μεταφορών και εξαθρολογισμό του κόστους. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλετε να πείτε σε σχέση με αυτό το θέμα. Έχουμε πολλές δυνατότητες ώστε να γίνουν οι σιδηροδρομικές ε, μεταφορές καλύτερες, αλλά όχι να κάνουμε και πιο ακριβές τις οδικές. Ο κύριος Ντελή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Εδώ είμαι, εδώ είμαι, εδώ μπροστά σας. Υπάρχουν θέματα τα οποία ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι για αυτά τα οποία λέτε στη μελέτη σας, καλά είναι, αλλά βλέπω ότι υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε μέτρα για να ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα. Στην ε, σελίδα 44 λέτε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να μειώσουν την κινητικότητα αντί να την κάνουν πιο καθαρή εντός παρενθέσεως. Ξέρετε ποιες είναι οι παρούσες τάσεις. Όταν εκπονήσετε το έγγραφό σας, βασιστήκατε σε μελέτες στις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά τη μείωση της κινητικότητας. Αν κάτσουμε όλοι στο σπίτι μας για μια εβδομάδα φερρυπίν, τι αντίκτυπο θα έχει αυτό ε, στο περιβάλλον. Υπάρχουν αριθμοί, υπάρχουν στοιχεία, αποδείξεις, επιστημονικές αποτελέσματα ή κάνουμε τα πρώτα δειλά τι σημαίνει η μείωση της κινητικότητας, κάτι το θετικό, θα υπάρχει θετικός αντίκτυπος ή πρόκειται για ένα νέο, κάτι το μοντέρνο πλέον στα μίδια. Σας ευχαριστούμε κύριε Ντελή. Βλέπετε πόσες πολλές ερωτήσεις και όλοι βεβαίως λέγουν ότι είναι μάλλον θετική η μελέτη σας, αλλά υπάρχει απεσιοδοξία και ερωτηματικά. Έχετε τέσσερα λεπτά για να κάνετε την απάντησή σας και να σεβαστούμε και το χρόνο που έχουν στην διάθεση τους οι διερμηνείς. Α, έχετε κάνει μελέτες, πρέπει να μπορείτε να μιλάτε και συνοπτικά. Καλά άκουσα. Έχω μόνο τρία λεπτά για να κάνουμε την ε, συζήτηση. Όσον αφορά ένα από τα θέματα που παρουσιάστηκαν είναι η πρόταση που κάναμε και κάποια από τα σχόλια είναι ότι μας προτείνεται κάτι πάρα πολύ καλό αλλά δεν είναι εφικτό, δεδομένου ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ πολύπλοκα. Αυτό το καταλαβαίνω. Και εγώ είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο και προσπαθώ να πω πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Αλλά στο τέλος βλέπω ότι υπάρχουν δυσκολίες στην εφαρμογή. Εγώ δεν έλαβα υπόψη το γεγονός ότι είναι τόσο δύσκολο να μπορέσει κανείς να διαπραγματευτεί με το Συμβούλιο ή να κάνει έναν ενιαίο οργανισμό όταν ε, οι διάφοροι τύποι μεταφορών είναι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους. Κάτι είπατε επίσης για την κινητικότητα και είπατε σε ποιο μέτρο λέμε ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι καλό. Επίσης, η μείωση της κινητικότητας, όπως είπε ο κύριος Ντέλη, είναι καλό ή μη καλό. Αυτές είναι οι προσωπικές απόψεις. Θα απαντήσω ως εξής. Η κινητικότητα αυξάνεται υπερβολικά, αλλά είναι και μέλος της ποιότητας της ζωής. Και τελικά το σημαντικό θέμα είναι να μπορέσει κανείς να βρει τη χρυσή τομή σε όλους τους τομείς ε, που επιτρέπουν να επιτύχει την βιωσιμότητα και την αηφορία. Και όπως ξέρουμε υπάρχει εδώ το κομμάτι το οικονομικό, το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό. Και μόνο έτσι και φτάνοντας στη χρυσή τομή θα μπορέσουμε να κάνουμε μία ισόρροπη ανάπτυξη η... αν η Ευρώπη δεν μπορέσει οικονομικά να αναπτυχθεί ισόρροπα, τι κατορθώνουμε. Η σωστή ισορροπία λοιπόν είναι η λύση. Και από αυτού θα πω ότι θα πρέπει τις επενδύσεις να τις δούμε διαφορετικά από το να έχουμε νέα αυτοκίνητα πιο οικολογικά τα οποία θα κυκλοφορούν στους δρόμους. Βεβαίω η μείωση τη ρήπανση είναι σημαντική, αλλά το κύριο θέμα για την κινητικότητα δεν είναι ο αριθμό των ε, υποδομών, αλλά το γεγονός ότι η κινητικότητα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ αναποτελεσματικό. Υπάρχουν νέες εξελίξει ε, στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται οι άνθρωποι, γιατί υπάρχει και η έλλειψη υποδομής. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις επενδύσεις ως έναν τρόπο για να διευκολύνουμε την ε, ε, σύνδεση και νομίζω με τον τρόπο αυτό ε, θα μπορέσουμε να διευκολύνουμε αυτό που και εσείς αναφέρατε, την ε, ηθική μετάβαση. Αυτό που παίζει ρόλο είναι να διευκολύνουμε και τα ηλεκτρικά οχήματα, να υπάρχουν ίση όρια ανταγωνισμού και με ρωτήσατε ποια ακριβώς είναι η γνώμη μου από αυτού. Και η γνώμη μου είναι ότι τώρα στην Ευρώπη ε, δεν υπάρχει ένα σύστημα ε, πρώτων βοηθειών και κατά τη δική μου άποψη αυτή η φορολογική προσέγγιση πρέπει να εστιάζεται σε περιβαλλοντικά θέματα. Και αυτός είναι ένας τρόπος ε, ίσων όρων ανταγωνισμού. Επίσης, τα κίνητρα, παραδείγματος χάρη, τα κίνητρα για να μοιράζει κανείς ένα αυτοκίνητο, να χρησιμοποιεί ε, πιο ε, καθαρά καύσιμα. Υπάρχει κατόπιν και ένα θέμα, το οποίο κατά την άποψή μου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και αφορά στο κατά πόσο είναι δυνατόν να περιοριστεί η κινητικότητα. Νομίζω ότι ανεξάρτητα από τα μέτρα τα οποία χρησιμοποιούμε, οι άνθρωποι θέλουν να μετακινούνται περισσότερο. Αυτά είναι, αυτό είναι στην πραγματική ζωή. Από την άλλη, αν οι άνθρωποι θέλουν να μετακινούνται, είναι διότι την ποιότητα ζωής τους ε, την εστιάζουν ε, στην κινητικότητα, στον ε, στο ότι θέλει κανείς να επισκεφτεί τη μητέρα του, άρα δηλαδή το να αναγκάζουμε τους ανθρώπους να μην μετακινούνται, αυτό δεν είναι αποτελεσματικό, γιατί πρέπει να σεβόμαστε την ελευθερία όλων. Σε τελική ανάλυση, ποιο είναι το καθοριστικό στοιχείο. Θα πρέπει να αγωνιστούμε ε, και ένα θέμα είναι η ευαισθητοποίηση, δηλαδή να, να εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους ε, και τα κίνητρα, κατά την άποψή μου, ε, οι εξωτερικοί παράγοντες ε, δεν λαμβάνονται υπόψη, δηλαδή ε, ταξιδεύουμε με ένα κόστος που είναι χαμηλότερο από αυτά που παράγουμε. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Ας προχωρήσουμε λοιπόν ε, σε κάποια άλλα στοιχεία. Και αναφέρατε επίσης το ότι πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και σε άλλα θέματα. Υπάρχει εδώ κάποια κριτική στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ένα από τα πράγματα που διαπιστώνουμε και ένα από τα πράγματα που υπάρχουν εδώ είναι σε ποιο βαθμό τα κονδύλια είναι αποτελεσματικά. Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε εργαλεία για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα. Επίσης, και αυτό είναι κάποια από τα θέματα που θέλω να δείξω, είναι σε ποιο βαθμό μπορούμε να έχουμε ένα μηχανισμό για να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα. Γιατί δεν είναι μόνο η οικονομική αποτελεσματικότητα, έχει και να κάνει με τις ισορροπίες. Αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των μεταφορών. Και εμείς ε, δουλεύουμε πάνω σε αυτό, ε, προσπαθούμε να αναπτύξουμε μηχανισμούς, αλλά πιστεύω ότι όσον αφορά το πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια, ε, πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω και σήμερα οι περισσότερες αξιολογήσεις που γίνονται γίνονται εστιάζονται κυρίως στα ε, διοικητικά θέματα και όχι τόσο στις ε, επιπτώσεις. Αυτό είναι ένας από τους λόγους γιατί και συστήνουμε να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο και ίσως ε, να αναπτύσσουμε και μία μέθοδο η οποία θα βοηθήσει έτσι ώστε να αποκομίσουμε μαθήματα για το μέλλον. Γιατί ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουμε είναι ότι δεν μπορέσαμε να μάθουμε πολλά από το παρελθόν για να τα εφαρμόσουμε για το μέλλον ευχαριστούμε. ευχαριστούμε, κύριε Βασάλο, για την παρουσίαση και τις απαντήσεις. Την επόμενη φορά θα δώσω χρόνο και στην κυρία Λάουρα Γαρίδο. Θέλετε να προσθέσετε κι εσείς κάτι? Για να συνοψίσετε πάρα πολύ γρήγορα. Το μόνο πράγμα το οποίο έρχεται στο μυαλό μου, γιατί μιλάμε για τον περιορισμό της ε, κινητικότητας, είναι η ε, καθημερινή ε, κινητικότητα. Δηλαδή, κατά πόσον πρέπει όλοι να πάμε σε ένα συγκεκριμένο χώρο για να εργαστούμε. Υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν και εάν ας πούμε πρέπει κανείς να πάει στη μητέρα του που είναι στο Παρίσι, δεν μπορώ να σας πω να μην πάτε με το αυτοκίνητο, αλλά Μπορείτε να μην πάτε με το δικό σας το αυτοκίνητο. Μπορείτε να πάρετε παραδείγματο χάρη το τρένο που σημαίνει ότι υπάρχουν ορισμένα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε έτσι ώστε πραγματικά να περιορίζουμε την κινητικότητα χωρίς ε, να αναγκάζουμε τους ανθρώπους να μην μετακινούνται όταν πρέπει να μετακινούνται. Αυτά απλό ήθελα να πω. Σε ευχαριστούμε για τη μελέτη, ευχαριστούμε τους διερμηνείς που έμειναν και μερικά λεπτά παραπάνω μαζί μας και ελπίζουμε ότι αυτά τα οποία είπατε θα εισακουστούν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο δικός χάρτης που έχει χαραχθεί ούτως ή άλλως είναι κάτι που πρέπει να τηρήσουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση. Και βεβαίως μεταφορές